Uh, good morning everybody. I think we're ready to start. Now our rapporteurs here. Καλημέρα. Είναι εδώ η συγητής μας για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Είναι ώρα λοιπόν να ξεκινήσουμε. Καλημέρα σας. Είναι η τελευταία μας συνεδρίαση πριν από τις καλοκαιρινέ διακοπές και νομίζω ότι τα μέλη της Επιτροπής μας ε, αξίζουν ε, τις καλοκαιρινέ διακοπές ε, με τη δουλειά που έχουν κάνει τους τελευταίους 7 μήνε. Έχουμε όμω πολλή δουλειά σήμερα και έχουμε και σημαντικές ψηφοφορίε. Χαίρομαι που είστε πολύ άριθμοι εδώ σήμερα. Θα ήθελα να αρχίσω τη δουλειά για την έκθεση Δίας Πρωτοβουλίας ε, που θα μας πάει μέχρι το δεύτερο ε, τμήμα του έτους. Είναι εδώ ο ε, Παύλος Αρίας Ετσεβερία να μας πει ορισμένα πράγματα πριν αρχίσει η συζήτηση και πριν ολοκληρώσουμε τη σχετική δουλειά πριν από το τέλος του έτους. Είναι μια σημαντική πράσινη βίβλος από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς για την ολοκληρωμένη αγορά δεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ολοκληρώνουμε αυτή τη δουλειά. Έχουμε την ε, κυρία ε, Σενέλοβα, τον κύριο Κρόιτσμαν, την κυρία Ρούλε, τον κύριο Μπίλαν ως σκιώδης εισηγητές. Δεν βλέπω κανέναν άλλον, είναι όμως πολύ ισχυρή ομάδα σκιωδών εισηγητών. Και έχουμε και τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ε, Εσωτερικής Αγοράς, τον αρμόδιο για το θέμα αυτό, ο οποίος είναι τακτικός επισκέπτης. Ε, μεταδιδόμαστε ζωντανά και στο διαδίκτυο. Φαντάζομαι ότι ε, πολλοί απασχολούμενοι στον τομέα θα παρακολουθήσουν τις συζητήσεις μας. Να ενημερώσω λοιπόν όσους μας παρακολουθούν ε, ζωντανά, να τους πω ότι υπάρχει και το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο για το οποίο, στο οποίο μπορείτε να ε, μας παρακολουθείτε σε μηνιαία βάση. Να δώσω το λόγο στον Παύλο Σαρία Ετσεβερία για να μας πει πώς βλέπει τα πράγματα σε σχέση με το θέμα αυτό και να ακούσουμε μετά και τα σχόλια των σκηδιωδών εισηγητών. Πρώτα ο Παύλο Αρίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίναμε ένα σημαντικό ψήφισμα κάτι το οποίο σημαίνει ότι είμαστε πραγματικά δεσμευμένοι για, μια, ε, για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μας υποστήριξαν όλες οι πολιτικές ομάδες και εγκρίναμε με ομοφωνία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις και τις πολιτικές ομάδες. Σήμερα το θέμα που μας απασχολεί είναι ύψης της σημασίας, διότι πρόκειται για έναν από τους βασικούς πυλώνες του ηλεκτρονικού εμπορίου για την αποστολή και την διανομή. Αυτό είναι, αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα πρέπει να έχουμε υπηρεσίες παράδοσης και διανομής υψηλής ποιότητας. Αυτό είναι ύψης της σημασίας για να προωθήσουμε τις πωλήσει μέσω διαδικτύου και να φτάσουμε στην ψηφιακή αγορά. Οι διαβουλεύσεις δείχνουν ότι έχουμε δύο βασικά προβλήματα. Από τη μία πλευρά δεν υπάρχει εμπιστοσύνη από τους καταναλωτές και ένα σύστημα το οποίο δεν τάσεται υπέρ των ΜΜΕ διασυνοριακά. Πολλοί καταναλωτές δεν αγοράζουν online, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για διασυνοριακή αγορά πολλοί Ευρωπαίοι καταναλωτές δεν δείχνουν εμπιστοσύνη και φοβούν, φοβούνται για τα προϊόντα που αγοράζουν μέσω διαδικτύου και γι' αυτό δεν τα αγοράζουν. Σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία του Green Paper της Επιτροπής, ο ένας στους δύο καταναλωτές, δηλαδή το 47%, δηλώνει ότι δεν αγοράζει online διότι δεν έχει εμπιστοσύνη φοβάται ότι δεν έχει επαρκείς πληροφορίες ή δεν θα του παραδοθεί το προϊόν. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση εάν θέλουμε να προωθήσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η ίδια η Επιτροπή θα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Είναι μία από τις πέντε προτεραιότητες για την επίτευξη της ενιαίας εσωτερικής αγοράς έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ βασικό ζήτημα για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις μας. Γι' αυτό και μία από τις βασικές προτεραιότητες είναι να ε, τονωθεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Γι' αυτό θα ορίσουμε έξι προτεραιότητες, ε, λεπτομερής πληροφόρηση του καταναλωτή για να ξέρει πότε θα του παραδοθεί το προϊόν, ποιο είναι το κόστος του, πώς πρέπει να το επιστρέψει αν δεν είναι ικανοποιημένος και ποιο θα ήταν το κόστος επιστροφής ο πολιτής στην ιστοσελίδα του, όπως προβλέπεται στη νέα οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή, όλα τα λεπτομερή στοιχεία κατά απλό και σαφή τρόπο. Επίσης, ευελιξία για την παράδοση και διαφοροποίηση των προσφορών. Ένας καταναλωτής μπορεί να διαπιστώσει ή να επιθυμήσει παράδοση λίγες μέρες μετά ή κάπου, ε, να παραδοθεί κάπου αλλού από την κατοικία του. Έτσι θα προωθήσουμε τις πωλήσει online και θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές και οι ΜΜΕ. Επίσης, ε, τάχιστη παράδοση. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθυστερήσεις έτσι ώστε οι αγορές online να είναι δελεαστικές. Τέταρτον, αποτελεσματικότητα. Ε, τα δέματα, τα πακέτα θα πρέπει να φτάνουν στο, στον προορισμό τους όποτε προβλέπεται. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν λογικές τιμές για τους καταναλωτές. Οι τηλεαγορές θα προωθηθούν εάν οι τιμές είναι δελεαστικές. Επίσης θα πρέπει να εξευρεθούν καινοτόμες λύσεις για τιμές που είναι πολλές φορές υπερβολικές. Έκτον, η παράδοση να μπορεί να γίνει ενδοκινοτικά ακόμα και σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές. Θα πρέπει οι καταναλωτές σε αυτές τις περιφέρειες να μπορούν να έχουν, να λαμβάνουν αυτά τα προϊόντα για αυτούς τους, ε, σε αυτές τις έξι προτεραιότητες θα πρέπει να, σταθούμε και αυτές τονίζουμε στην έκθεση. Η άλλη προτεραιότητα σχετίζεται με τις ΜΜΕ. Κατά την άποψή μου θα πρέπει η εσωτερική ψηφιακή αγορά να ε, προωθήσει τη δραστηριότητα των ΜΜΕ πολλές φορές η διασυνοριακή παράδοση ε, έχει ένα υψηλό κόστος και δεν συμφέρει η πώληση. Πολλές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα και δεν υπάρχει εναρμόνιση. Ως προς τη σήμανση, τους ε, ταχυδρομικούς κώδικες, την ε, συσκευασία κλπ. Θα πρέπει να λήξει αυτή η ασύμφορη κατάσταση και γι' αυτό μιλήσαμε και για την προσβασιμότητα των ΜΜΕ της ψηφιακής αγοράς, διότι αποτελούν το 99% των επιχειρήσεών μας και οδηγούν σε ε, πολύ υψηλές αποδόσεις. Θα πρέπει οι ΜΜΕ να μπορέσουν να ανταγωνιστούν με ίσους όρους. Όταν, μιλάμε, όταν μιλήσαμε για το ψήφισμα ηλεκτρονικού εμπορίου, μιλούσαμε για ΜΜΕ συν ψηφιακή οικονομία που οδηγεί στην ανάπτυξη. Αυτή η εξίσωση ισχύει και για τις υπηρεσίες αποστολής. Θα πρέπει να υπάρχουν πραγματικές ε, υπηρεσίες αποστολής της αποστολής με λογικές τιμές έτσι ώστε να μπορέσουν οι ΜΜΕ να ανταγωνιστούν τους γίγαντες του ίντερνετ. Αυτό θέλουμε να το προωθήσουμε. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ε, έχουν βελτιώσεις, να υπάρχει δηλαδή διαφάνεια ως προς τις υπηρεσίες και προσβασιμότητα σε καλύτερη προσφορά σε καλύτερες προσφορές. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει εποπτεία από τους αρμόδιους οργανισμούς έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και προσβασιμότητα έτσι ώστε να μην υπάρξουν καταχρήσεις. Επίσης, τυποποίηση των διαφόρων διαδικασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί πολλές φορές οι ΜΜΕ δεν μπορούν να ανταγωνιστούν διασυνοριακά. Δεν υπάρχουν τυποποιημένες σημάνσεις ε, των ταχυδρομικών ε, κωδίκων και των κωδικών ασφαλείας. Ιδιαίτερα όσον αφορά την ανιχνευσιμότητα όπου το σύστημα διαφέρει από κράτος σε κράτος. Θα πρέπει να ενοποιήσουμε αυτές τις διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να μειωθεί το, το επιπρόσθετο κόστος, να υπάρξουν πλατφόρμες ανταλλαγής πληροφοριών για να βελτιωθεί η κατάσταση και για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, διότι έτσι μόνο θα μπορέσει να ανταποκριθεί η βιομηχανία χωρίς να υπάρξουν στρεβλώσεις αγορών που πολλές φορές ε, αποτελούν μεγάλο πονοκέφαλο για τον νομοθέτη. Θα πρέπει να φτάσουμε σε καλύτερη απόδοση μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας της βιομηχανίας και να φτάσουμε σε νέες πρακτικές. Νομίζω ότι είμαι, μάλλον είμαι πεπισμένος ότι έτσι θα φτάσουμε σε μια καλύτερη ανταπόκριση. Θεωρώ επίσης η ύψη της σημασίας ώστε τα θεσμικά όργανα να ελέγξουν διεξοδικά την ισχύουσα ρύθμιση και νομοθετικό πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε πολιτικές που θα προωθήσουν τις άνοφοι πολιτικές. Παράλληλα θα πρέπει να διενεργηθούν μελέτες για να δούμε κατά πόσο είναι η διαφανής ο τομέας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πληροφορίες έτσι ώστε να πρέπει να αλλάξουμε το τρέχον ρυθμιστικό πλαίσιο και πολλές φορές θα πρέπει να προωθήσουμε πολιτικές έτσι ώστε να φτάσουμε στην τυποποίηση των διαφόρων διαδικασιών για να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση και διαφάνεια του τομέα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, η οδηγία για τις τηλεαγορές, η οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή μιλά για διεξοδικές ε, πληροφορίες και εμπιστοσύνη του καταναλωτή για τις προθεσμίες, το κόστος κλπ. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επίτροπη να εφαρμόσει αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο. Επίσης, δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις λόγω ε, Δηλαδή, όπως είδαμε πολλές φορές σε διάφορες μελέτες, οι απομακρυσμένες περιοχές δεν καλύπτονται. Η οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ε, έληξε πέρσι ως προς την ε, προθεσμία μεταφοράς και βλέπουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε με την ενιαία ψηφιακή αγορά, λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη ψηφιακή επανάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει διεξοδική μελέτη. Χρειαζόμαστε επίσης ε, πληροφορίες για το πραγματικό κόστος της παροχής υπηρεσιών, ε, έτσι ώστε να δούμε ποια είναι τα κενά της αγοράς ή άλλες πληροφορίες Νομίζω ότι θα πρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα τις αναθεωρήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ε, πλήρες πληροφορίες. Αυτά είναι ορισμένα από τα μέτρα που θα πρέπει να προωθήσουμε εδώ για να φτάσουμε σε μία έννοια ψηφιακή αγορά υπηρεσιών ε, αποστολής. Θα πρέπει να υπηρετούμε πάντα τον καταναλωτή και της ΜΜΕ. Είμαι πεπισμένος ότι οι συνάδελφοι, οι σκιώδεις και οι άλλες πολιτικές ομάδες έχουν συγκεκριμένες ιδέες που θα προωθήσουν και θέλω να τους ακούσω. Θα πρέπει να προωθήσουμε αυτό τον διάλογο και γι' αυτό θα ήθελα να μου διαβιβάσουν προτάσεις για βελτίωση. Όχι μόνο εδώ, αλλά στις ξεχωριστές συνεδριάσεις που θα προωθήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να προωθήσουμε μία πραγματικά καρποφόρα συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο, για όλα αυτά που μας είπες. Θα είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα, ενδιαφέρον αυτό το εγχείριο, εγχείρημα. Να δώσω τώρα το λόγο στους σκιώδεις συζητητές, η κυρία Σενέλοβα πρώτα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε μιλήσω για την πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μαζικά οι καταναλωτές και αυτή η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είχε ως σκοπό την ενιαία αγορά και σε ό,τι αφορά θέματα επιμελητίας, σε ό,τι αφορά θέματα πωλήσεων. Πρόκειται για μια πολύ δυναμική, αν θέλετε, αγορά της οποίας το δυναμικό θα πρέπει πλήρως να αξιοποιήσουμε. Το ίμιση των καταναλωτών δηλώνει ότι φοβάται να κάνει αγορές μέσω του διαδικτύου. Γιατί φοβούνται. Για τον καταναλωτή είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστούν και τέτοια προβλήματα σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι πολίτες και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν ε, ε, βρίσκονται σε άλλη χώρα θεωρούν ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θεωρώ ότι δύο βασικοί όροι θα πρέπει να ε, συνδράμουν για την άρση των εμποδίων. Καταρχάς, ποιότητα των υπηρεσιών. Αυτό το απαιτεί ο καταναλωτής να φτάσει το προϊόν σε αυτόν με άρεστες συνθήκες, με διαφάνεια και επιθυμεί επίσης ο καταναλωτής να έχει δικαίωμα επιστροφής ε, του προϊόντος και μάλιστα με σαφείς όρους. Για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτή η ποιότητα για την αποστολή των πακέτων. Θα ήθελα να αναφέρω και κάποια σχετικά μέτρα τώρα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει εγγύηση για την αποστολή του πακέτου. Την ευθύνη αυτή θα πρέπει να την διευκρινίζουν και την αναλαμβάνουν σε κάθε περίπτωση ο πολιτής και ο διανομέας. Και για την διευκόλυνση της βασικής επικοινωνίας μεταξύ του ε, εμπόρου και του καταναλωτή είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οι καταναλωτές βασικά απαιτούν πρακτικές λύσεις επί των οποίων θα μπορούν να συμφωνήσουν με τους πολιτές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και ένα κανάλι επικοινωνίας χωρίς ε, χρέωση. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί και η πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες παραγγελίας στην ύπνες ε, ε, περιοχές. Επίσης, βασικό είναι το δικαίωμα επιστροφής και οι πληροφορίες για την αποστολή. Από τεχνικής άποψης, είναι απαραίτητο όλοι οι συμμετέχοντες να φροντίσουν για την ταυτοποίηση των πακέτων και μάλιστα από την αρχή της αποστολής του μέχρι το τέλος της παράδοσής τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επιστροφές, θεωρώ ότι καλό είναι να υπάρχει ένας τυποποιημένος κώδικας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση επιστροφών θα πρέπει να υπάρχει ένα εύρυθμα, ένα εύρυθμο σύστημα. Θεωρώ ότι η εφαρμογή της οδηγίας θα μπορούσε να βοηθήσει και προς αυτή την κατεύθυνση. Και σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Στον τομέα αυτό ασφαλώς θα πρέπει να αντίθεται προτεραιότητες και συνθήκες και όροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημαντικά είναι τα συστήματα ADR και ODR. Αλλά σε ό,τι αφορά την αποστολή πακέτων θα πρέπει να το θεωρήσουμε αυτό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις εργασιακές συνθήκες των υπαλλήλων. Αυτό σε όλη την αλυσίδα αποστολής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα ήθελα να πω ότι το όριο των 30 κιλών, το οποίο αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί μεγάλο πρόβλημα γιατί ε, δεν συνάδει με την εργασιακή νομοθεσία, το εργατικό δικαίο πολλών κρατών μελών. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο καταναλωτής σε πολλές περιπτώσεις αποφεύγει να αγοράσει μέσω διαδικτύου κάποιο προϊόν λόγω της τιμής αποστολής. η οποία σήμερα επιβαρύνεται και από το διοικητικό κόστος. Εγώ τι να πω. Βλέπω ότι υπάρχει κάπως ένας παραλληλισμός, αν θέλετε, και με τα τέλη περιαγωγής. Δεν είναι δυνατόν σε μια πραγματικά ενιαία αγορά να υπάρχουν τέτοια χρέη να υπάρχουν τέτοια τέλη. Τέλος, να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πότε θα μας διαθέσει τα αποτελέσματα της δημόσιας ακρόασης. Είχατε πει ότι θα μας τα διαθέσετε στις αρχές του έτους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σίγητα για την συνεργασία. Good. Thank you very much indeed. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Κρότσμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. διαπιστώνουμε επανειλημμένα ότι στην εσωτερική αγορά ε, δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση σε διασυνοριακό επίπεδο. 9% μόνο κάνουν τις αγορές. 1% στο Λουξεμβούργο, μόνο 1% στη Ρουμανία, 35% στο Λουξεμβούργο. Δηλαδή υπάρχει τεράστιο δυναμικό βελτίωσης και διαπιστώνουμε επανειλημμένα ότι ένα βασικό θέμα για την αποστολή των πακέτων διασυνοριακά μάλλον ότι η αποστολή των πακέτων διασυνοριακά αποτελεί ένα από αυτά τα εμπόδια και το σχετικό κόστος. Αυτό αποτελεί ένα μόνο κομμάτι του προβλήματος. Πέρα από την ανασφάλεια για την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή, όλα αυτά δεν είναι πάρα πολύ σαφή στο ηλεκτρονικό εμπόριο και πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρούν ότι δεν είναι αρκετά ελκυστικό το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αναφέρει αυτά στην Πράσινη Βίβλο και αναφέρει ε, θέματα αποστολής πακέτων. Είναι απαραίτητο να ληφθούν κάποια μέτρα, τα οποία όμως σε πολλές περιπτώσεις είναι αμφισβητήσιμα. Η πιο μεγάλη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την αποστολή των πακέτων, των όρων ε, αποστολής θεωρούμε ότι θα ήταν πολύ καλό να υπάρχει και να διευκρινίζεται σε μια αρχική σελίδα ακόμα στα εσείς σελίδες, προκειμένου να υπάρχει και διεύρυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Κάποιες ε, υποχρεωτικές ε, ρυθμίσεις θεωρούμε ωστόσο ότι δεν θα πρέπει να επιβληθούν, γιατί θεωρούμε ότι υπονομεύουν τα δικαιώματα του καταναλωτή. Οποιαδήποτε ρύθμιση θα πρέπει να επαφίεται στα χέρια των εμπόρων και των καταναλωτών και των δύο. Τα χαμηλά περιθώρια κέρδου, υποδεικνύουν ότι ο ανταγωνισμό λειτουργεί καλά. Τα μέτρα αυτά σε ό,τι αφορά το κόστος τη αποστολή, είναι δύσκολο να εφαρμοστούν γιατί δεν υπάρχουν τιμέ στι αγορές και τα αναγκαστικά πλαφών στις τιμές ενδεχομένω να διώξουν από την αγορά κάποιους ε, εμπόρους. Κοιτάξτε, αναφέρομαι σε κάποια κριτικά σημεία, κρίσιμα σημεία της πράσινης βίβλου, με τα οποία δεν συμφωνούμε γιατί θεωρώ ότι θα ήταν αντιπαραγωγικά. Θεωρώ ότι πολύ απλά ο καταναλωτής θα πρέπει να αποφασίσει ποιε προσφορέ θέλει να δεχτεί και ποιε δεν θέλει να δεχτεί. Και δεν είναι, είναι αρμοδιότητα να προδιαγράψει όρους που θα είναι αντιπαραγωγικοί και θα είναι αντίθετα και με το πνεύμα της αγοράς, γιατί πολλά τα οποία ορίζουμε στην πραγματικότητα δεν προωθούν την αγορά. Γι' αυτό λοιπόν ανέφερα τα βασικά σημεία της πράσινης Λίγου με τα οποία δεν συμφωνώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, η κυρία Ρούλα μου προκαλεί μεγάλη έκπληξη, αλλά συμφωνώ μαζί σας κύριε Κρότσμαν σε κάποιους ε, τομείς. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι είναι πιο σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια παρά η απόπειρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ρίξει το κόστος. Κοιτώντα τι γίνεται ε, στην τομέα, κοιτώντα ε, τι διαφορές υπάρχουν στους μισθούς, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και το πρόβλημα μου και η εντύπωσή μου είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μεγάλη πίεση χρόνου στους ανθρώπους αυτούς και αντίστοιχα μεγάλο είναι το ποσοστό σφάλματος. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και στα ταχυδρομεία είναι μεγάλο το ποσοστό σφάλματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό ο καταναλωτής να μπορεί να ε, επιλέγει αυτός και να επηρεάζει αυτός την παροχή υπηρεσιών, γιατί υπάρχουν μεγάλες διάφορες. Ε, εγώ Για παράδειγμα, θα ήθελα ε, να μπορούν να παραδίδονται τα πακέτα σε ώρε μη εργάσιμε και αυτό φαντάζομαι ισχύει για τον πιο πολύ κόσμο. Όταν λοιπόν παραγγέλνω ένα πακέτο, πώ θα μπορέσουν να το παραλάβω. Αυτό, α πούμε, καλό θα ήταν να ρυθμίζεται ελεύθερα, ιδιαίτερα στο διασυνοριακό εμπόριο. Πώς παραδίδονται λοιπόν τα πακέτα όταν κανείς δεν είναι στο σπίτι. Η διαφάνεια θεωρώ ότι είναι το βασικό στοιχείο και προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε. Αλλά όπως και ο εισηγητής δεν θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη νομοθετικής ε, πρότασης. Αυτό που χρειάζεται είναι να εφαρμοστούν πιο σωστά και να ελεγχθούν οι ήδη υφιστάμενες νομοθεσίες. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάιντι. Θα ήθελα να σας ζητήσω λίγη ησυχία να κάνετε, ειδικά όταν μιλούν ε, οι ομιλητές. Είναι χαμηλοτάβανη η αίθουσα εδώ και μερικές φορές είναι λίγο δύσκολο. Ακούγονται πάρα πολύ ε, οι άλλες ομιλίες ε, πριν από την ψηφοφορία. Αν θέλετε να κάνετε συζητήσεις, παρακαλώ, εκτός της αίθουσας. Ο Άνταμ Μπίλαν. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο? Άνταμ Μπίλαν και μετά θα δώσω το λόγο ε, στην, Γενική Διεύθυνση Ιστορικής Αγοράς. Τρία βασικά ζητήματα θίγονται για τους καταναλωτές κατά τις ηλεκτρονικές αγορές τους. Πώς μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική ε, η αγορά ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η σχέση κόστους και ωφέλου, πώ είναι δυνατόν να είναι καλύτερη και πώ είναι δυνατόν να είναι καλύτερες οι επιλογές για τους καταναλωτές. Πώς μπορεί κανείς επίση να ενισχύσει τη διαδραστικότητα μεταξύ των διαδικασιών παράδοσης ε, από τους διάφορους φορείς και τους ε, χειριστές τη παράδοση αυτή. Πριν ε, δούμε λύσεις για να καταστεί πιο αποτελεσματική παράδοση, πρέπει να σκεφτούμε την αγορά που είναι πολύ νέα, πολύ δυναμική και σύμφωνα με εκτιμήσεις κατά τα επόμενα 10 έτη ο όγκος παραδοσιακών γραμμάτων θα περιοριστεί κατά 10 με 20% που σημαίνει ότι το ηλεκτρονικό ε, εμπόριο και το, ε, τα ηλεκτρονικά δέματα θα αποτελέσουν σημαντικό τμήμα τις δραστηριότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να γίνουν συνεπώς πιο ανταγωνιστικές και πιο αποτελεσματικές. Βέβαια, οι διασυνοριακές συναλλαγές ε, ε, είναι λιγότερες από τις παραδοσιακές ε, εγχώριες. Μερικές φορές υπάρχει ένα γλωσσικό εμπόδιο, για παράδειγμα, και δεν υπάρχει καμιά νομοθεσία που να μπορεί να βοηθήσει ως προς αυτό μερικές φορές, εξαρτάται από τις μεμονωμένες αγορές ε, των κρατών μελών, μερικές φορές διασυνοριακές ε, συναλλαγές ηλεκτρονικές όντως λαμβάνουν χώρα. Υπάρχουν επίσης φορολογικά ζητήματα. Όταν λοιπόν προσπαθεί κανείς να καταστήσει πιο αποτελεσματική και πιο ανταγωνιστική την αγορά, πρέπει να το εξετάζει όχι μόνο από την άποψη του τελικού χρήστη της μικρομεσαίας επιχείρησης, αλλά και του πολιτή, δηλαδή των εταιριών συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και σε αυτή την περίπτωση αν ας πούμε κάποιος δεν θέλει να κάνει διασυνοριακή αγορά ηλεκτρονικός γιατί δεν ξέρει τη γλώσσα, ε, μπορεί κάποιε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να θέλουν μόνο ε, εντός μιας χώρα να δραστηριοποιηθούν. Πρέπει να σεβαστούμε αυτή την επιλογή. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι αυτή η ιδέα των ηλεκτρονικών, ε, τη ηλεκτρονική αγορά δεμάτων, αλλά είναι πολλά που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να έχουμε ηλεκτρονικέ μηχανέ. Μπορεί πούμε, να μπορεί κάποιο να, να, να, παραλάβει το δέμα του σε ε, ένα βενζινάδικο. Υπάρχουν πολλά μειονεκτήματα σήμερα, γιατί αναπτύσσεται πολύ γρήγορα αυτή η αγορά, οπότε αν θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, τώρα είναι η στιγμή να το κάνουμε. Ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιες είναι οι επιλογές και σχέση με την ε, ανταγωνιστικότητα και τις καλύτερες τιμές για τους ε, καταναλωτές. Γιατί το αναφέρεται αυτό στη πράσινη βιβλίο και δεν μπορώ να φανταστώ τέτοιου είδους λύσεις χωρίς ισχυρή, ισχυρή παρέμβαση στην αγορά. Ευχαριστώ. Πρόεδρο. ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και τους σχεδόν ε, εισηγητές να... να δώσω το λόγο στον ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Φόξ, δεν βλέπω τίποτα. Μήπως μπορείτε να πάτε λίγο πιο εκεί για να τον βλέπω. Προσπαθώ να του μιλήσω και να του δώσω το λόγο. Βέρνενστάιν, να σου δώσω το λόγο. Να πω κάτι γενικότερο. Πέρσι τον Νοέμβριο λάβαμε την πράσινη βίβλο. Κάναμε λίγο, λίγο, λίγο, πέρσι λίγος χρόνος μέχρι να ε, ασχοληθούμε με αυτήν. Όχι επειδή δεν θέλαμε, αλλά επειδή είχαμε και άλλα πολλά πράγματα να κάνουμε. Θα μας ενδιαφέρει, όπως είπε και η κυρία Σενελόβα, να μας πείτε Συγγνώμη, μήπως μπορείτε να καθίσετε, επαναλαμβάνω, δεν βλέπω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε νέα από τις διαβουλεύσεις που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί σας και να μας ενημερώσετε έτσι, να σας δώσω το λόγο για να σχολιάσετε που βρισκόμαστε στις συζητήσεις, δεδομένου ότι έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που ε, δημοσιεύσατε την ε, πράσινη βιβλίο. Ναι, ευχαριστώ Μάλκολ, Πάμπλο και τους υπόλοιπους ε, ομιλητές. Να αρχίσω με το θέμα του χρονοδιαγράμματος, το οποίο το ανέφερες Μάλκομ στο τέλος. Ναι, έχει περάσει χρόνος ανάμεσα στην δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου. 180 ε, απαντήσεις λάβαμε. Μας πήρε πολύ χρόνο να εξετάσουμε όλο αυτό το υλικό, να το συζητήσουμε με τους ενδιαφερόμενους φορείς όταν χρειάστηκαν περισσότερες ε, διευκρινήσεις, ε, είχαμε πολλά εργαστήρια, πολλέ διμερεί, πολυμερεί συναντήσει για να αξιολογήσουμε αυτά που είχαμε δει και αυτά που είχαμε μάθει. Είμαστε πεπισμένοι ότι ναι, η ταχύτητα είναι πάντα σημαντική, αλλά δεν θέλουμε να είμαστε επιπόλαιοι στι λύσεις που θα προτείνουμε, γιατί κάποιε από τους ομιλητέ είπαν ότι είναι ένα πολύ περίπλοκο περιβάλλον που αλλάζει ραχδαία και το τελευταίο πράγμα που θα θέλαμε ήταν να φτάσουμε σε ταχύτατες ε, υπερβολικές ε, λύσεις. Ελπίζουμε μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη να έχετε κάποιον χάρτη πορείας, ε, σχέδιο δράσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά τις διαβουλεύσεις για την Πράσινη Βίβλο, σε μεγάλο βαθμό συμφωνούν ως προς την ανάλυση τους. Όπως ακούσαμε και από τις παρεμβάσεις εδώ σήμερα, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη συνένεση όταν πρόκειται να βρούμε λύση, κάτι το οποίο ακούσαμε και στη σημερινή συζήτηση. Η ανάλυση, για την ανάλυση τώρα υπήρχε ευρεία συμφωνία. Όταν άκουσα το Πάμπλο να αναφέρει την ουσία του σχεδίου έκθεσής του, συνάδει πλήρως με αυτά τα οποία διαπιστώσαμε κι εμείς, κάτι το οποίο πραγματικά μας παρηγορεί. Όντως, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυξάνεται ραγδαία, όλες οι μελέτες, έρευνες, στατιστικές το επιβεβαιώνουν. Ένα ακόμη στοιχείο να σας αναφέρω που δεν το έχουμε πει ως τώρα. Η Copenhagen Economics την έκανε αυτή τη μελέτη για μας. Σε ποιο βαθμό, κάποιες, πόσες συναλλαγές στο διαδίκτυο σταματούν λόγω της παράδοσης Πάει κάποιος ας πούμε στο ίντερνετ, βρίσκει τα αγαθά που θέλει, αλλά επειδή ανησυχούν για τα θέματα της παράδοσης, 68% εγκαταλείπουν τη συναλλαγή αυτή. Αυτό το οποίο δείχνει ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό για όλους, όχι μόνο για τον καταναλωτή, αλλά και για τους ε, λιανοπολιτές, ε, για τους υπεύθυνους παράδοσης που έχουν τη δυνατότητα να παραδώσουν ε, ε, τα ε, δέματα αυτά, τα αγαθά αυτά. Όσον αφορά τώρα τους στόχους, συμφωνώ με αυτά που είπε ο Παύλο. Οι υπηρεσίες ε, σε καλές τιμές, υψηλής ποιότητας, διασυνοριακές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσβασιμότητα και στις περιοχές της υπαίθρου και στις περιφέρειες της Ευρώπης που είναι λιγότερο ανεπτυγμένες ως προς την, το ηλεκτρικονικό εμπόριο. Όντω, μπορεί λοιπόν να δώσει πολλές λύσεις αυτή η προσπάθεια και ειδικότερα για όλους όσους ε, δεν θα ήταν ε, ο βασικός στόχος αυτής της προσπάθειας. Συμφωνώ λοιπόν απολύτω με όλα όσα είπε ο Παύλο, συνάδει πλήρω με τη συλλογιστική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτον, χρειαζόμαστε Υπηρεσίε που ανταποκρίνονται στι ανάγκε των λιανοπολιτών και των καταναλωτών. Οι καταναλωτέ θέλουν να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα δέματά του και οι πολιτέ το ίδιο. Χρειαζόμαστε πολύ καλύτερες λύσεις, αποτελεσματικέ διαδικασίε, Όλοι συμφώνησαν σε αυτό. Και για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, κάποιο το είπε αυτό στο τέλο, ο κύριο Μπίλαν νομίζω, χρειαζόμαστε πιο ευθυγραμμισμένε αποτελεσματικέ διαδικασίε. Γι' αυτό αυτή η διάσταση τη ε, διαδραστικότητα είναι πάρα πολύ ισχυρή στην πράσινη βίβλο. Πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να συνεργαζόμαστε καλύτερα ο ένας με τον άλλο. Κατά τη γνώμη μας αυτό δεν είναι επιβλαβές για τον ταχυδρόμο, ο οποίος θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, αν υπάρχουν ε, πλεονεκτήματα ως προς τις τιμές για τον τελικό καταναλωτή και αν κάποια στιγμή όλοι οι φορείς ε, πρέπει δύο-τρεις φορές να βάλουν ετικέτες, αυτό θα στοιχήσει πολλά λεφτά χωρίς να είναι υποφελές για κανέναν. Οπότε υπάρχουν πολλά στοιχεία στο σύστημα που μπορούν να βελτιωθούν για τη μείωση του κόστους. Κυρία Σενέλοβα, Αναφερθήκατε συγκεκριμένα στις ε, συνθήκες εργασίας και στην απασχόληση, όπως ε, είδατε στην πράσινη βίβλο. Αναφέρουμε την ιδέα της αηφορίας, κάτι το οποίο είναι σημαντικό για μας. Θέλουμε αποτελεσματικές διαδικασίες, ε, όμως θέλουμε και κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες να λαμβάνονται υπόψη. Δεν θέλουμε ο να πληρώσει την ύφη για όλα αυτά. Ο προγραμματισμός είναι πολύ σημαντική πτυχή. Οπότε όταν όλα αυτά δρομολογούνται, υπάρχουν νέες ε, ε, υπηρεσίες, νέα προϊόντα, όλη αυτή η πτυχή της αηφορίας θέλουμε να ληφθεί υπόψη. Κύριε Κρόιτσμαν, αναφερθήκατε σε αυτά τα τμήματα της Πράσινης Βίβλου που αναφέρονται σε πιθανές, παρεμβάσει πιθανές παρεμβάσεις ε, στην αγορά, δηλαδή ανώτατα όρια τιμών κλπ. Μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι η πράσινη βίβλος ε, σκοπό είχε να διερευνήσει ένα πλήρες φάσμα επιλογών, να δει τι πιστεύουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για το θέμα αυτό και μπορώ να σας πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ενδιαφερομένων φορέων δεν θα ήθελαν υπερβολική ρύθμιση σε αυτή τη φάση, ούτε και εμείς θέλουμε. Μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό σε τρεις ε, χρόνια και να πούμε ότι έχει εξελιχθεί η αγορά και να δούμε ε, ότι ε, τότε πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα, να βελτιώσουμε τα πράγματα. Όσοι άλλως στο χάρτη πορείας μας θα υπάρχει η ρήτρα αναθεώρησης, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος υπερβολικά τώρα να παρέμβουμε σε, αυτά τα, αυτές τις πιο ανώριμες αγορές. Μπορώ λοιπόν να σας καθησυχάσω προς αυτό. Κυρία Ρούλε, είπατε ότι η διαφάνεια είναι πιο σημαντική από την τιμή. Για μας η διαφάνεια είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες, πληροφορία και διαφάνεια να ακούσαμε αυτό και από τους ομιλητές, ενημέρωση για τους καταναλωτές, να γνωρίζει ο καταναλωτές ε, τι μπορεί να περιμένει, να ξέρει ο καταναλωτής τι επιλογές έχει αν θέλει να αγοράσει κάτι διασυνοριακά. Όμως και η διαφάνεια που πολύ έξι μόνο αναφέρατε, για τους ρυθμιστές, ε, για τις αρχές να μπορούν να καταλάβουν πλήρως αυτά τα δια, αυτές διασυνορικές αγορές για τα δέματα που είναι πολύ αδιαφανείς για την ώρα. Αν θέλουμε να δώσουμε στις αγορές μια δυνατότητα να βελτιωθούν, να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, χρειαζόμαστε ε, εξασφάλιση του ότι οι δημόσιες υπηρεσίες ε, στα κράτη-μέλη για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρουμε κατά πόσο, ξέρει εάν έχουν γίνει σεβαστοί οι κανόνες, πρέπει να μπορεί να επιβλέπει και να παρακολουθεί την κατάστασή τους. Όσον αφορά τώρα τις τιμές. Πρώτον, θέλουμε να βελτιώσουμε, να μειώσουμε το κόστος και ελπίζουμε ότι αυτό θα σημαίνει και μείωση των τιμών αλλά το κόστος πρέπει να μειωθεί όπως είπα προηγουμένως και ειδικότερα ως προς τις διασυνοριακές τιμές ε, μεγαλύτερες ε, διαδικασίες σημαντικότερες ε, διαδικασίες ευθυγράμμισης μπορεί να σημαίνουν μείωση του κόστου σημαντική. Ο κύριος Μπίλαν είπε επίση ότι οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές δεν θέλουν τα, δύο, δεν δεν θέλουν τα ίδια πράγματα. Δίκιο έχετε σε αυτό. Δεν θέλω να υποχρεώσω κανέναν να αγοράσει κάτι διασυνοριακά, ούτε θέλω ένα ε, τυποποιημένο προϊόν να το, να το επιβάλλω σε κάποιον. Ε, πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα επιλογής. Αν κάποιος θέλει μια πολύ φθηνή παράδοση και δεν έχει σημασία πόσο ε, θα αργήσει να έρθει το δέμα του, πρέπει να μπορούμε να του δώσουμε αυτή την επιλογή. Αν κάποιος βιάζεται, πρέπει και αυτός να έχει αυτή την επιλογή δεν είναι δυνατόν να έχουμε μία λύση για όλους. Και φυσικά όχι μέσω άκαμπτης νομοθεσίας. Νομίζω ότι αυτό συνοψίζει ε, τα περισσότερα από υπόθηκαν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ καλή ευκαιρία εκκίνησης. Παύλο, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλεις ε, να μας μιλήσεις για το χρονοδιάγραμμα και να συνοψίσεις κάπως. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χειώδεις, τους ηγητές και την Επιτροπή. Η εργασία θα είναι ιδιαίτερα καρποφόρα. Το Σεπτέμβριο δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ως προς το χρονοδιάγραμμά μας, Πρόεδρε, θα το δούμε, μπορούμε να το δούμε, να δούμε τις ε, προθεσμίες και για το Σεπτέμβρη. Τώρα, στις 26 Αυγούστου τροπολογίες, 25-26 στο ΙΜΚΟ, προθεσμίες 8 ε, Οκτωβρίου και στις 4-5 Νοεμβρίου θα ψηφιστεί για τις τροπολογίες συμβιβασμών 27-28 Νοεμβρίου και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 17 ε, ε, Δεκεμβρίου, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ε, ευχόμαστε ένα παραγωγικό καλοκαίρι στη σύνταξη της έκθεσης και θα επανέλθουμε. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους όσους προσήλθαν για την ψηφοφορία. Ε, χτες η αίθουσα δεν κλιματιζόταν, γι' αυτό μπορείτε να βγάλετε και τα σακάκια σας, αν το επιθυμείτε. Εάν το θέλετε, αν θέλετε να το κάνετε μπορείτε. Ακολουθήστε τον πρόεδρο. Uh, so we have some serious work to do Λοιπόν, πολύ σοβαρή εργασία Ο κύριος ε, Τόνι Μπλερ, ο οποίος ε, πάντα έβγαζε το σακάκι στην αρχή της συνεδρίασης, είναι ο πρώην πρωθυπουργός τον οποίο ακολουθώ. τα γράμμα. Λοιπόν, καθίστε. θα ήθελα να κάνω ορισμένες ανακοινώσεις και να σας μιλήσω για ορισμένα θέματα που δεν είναι υποψηφοφορία. Βλέπω ότι ο Μάρκ Ταραμπέλα και ο Φιλίπ και Ζουβέ είναι παρόντες. Θέλαμε να ψηφίσουμε, σας παρακαλώ, ησυχία. Σας λέω σημαντικά πράγματα. Σήμερα θέλαμε ε, στο τομέα των δημοσίων συμβάσεων να επικυρώσουμε την εργασία του Συμβουλίου. Πρόκειται για ε, δύσβατα και πολυσχηδή ζητήματα. Ήταν πολύ δύσκολο να δούμε όλα τα νομοθετήματα. Τελειώσαμε με αυτή την εργασία και αύριο θα εγκριθούν από το Συμβούλιο. Και μετά θα έχουμε μία επίσημη επιστολή την επόμενη εβδομάδα, από όσο γνωρίζω. Δεν είχαμε επίσημη έγκριση της Κορεπέρ σήμερα και μετά θα λάβω την επιστολή, άρα θα ψηφίσουμε το Σεπτέμβριο με την πρώτη ευκαιρία. Αυτά περί αυτού. Τώρα, ως προς την πρόταση όπου ήμασταν επιτυχείς για ε, θέματα που αφορούν την Πενεντέτ Βενιόν, της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε με ένα πολύ σημαντικό θέμα, όχι μόνο για την απασχόληση και ανταγωνιστικότητα της εσωτερικής αγοράς, αλλά και ως προς τα δικαιώματα του πολίτη, θεμελιώδη δικαιώματα ως προς την κινητικότητα. τάχει θα ήθελα να σας πω ότι οφείλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν, ιδιαίτερα τους σκιώδεις. Θεωρώ ότι ήταν ανέλπιστο αυτό το αποτέλεσμα. Είχαμε αγαστή συνεργασία μεταξύ τριών θεσμικών οργάνων και σας ευχαριστώ γιατί παρακολουθείτε τις εργασίες εδώ και τρία χρόνια, δύο χρόνια. Μπορέσατε να ανταποκριθείτε και βοηθήσατε και τις διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ιρλανδική Προεδρία είναι παρούσα. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω όμως διότι μας ε, συνέδραμε ιδιαίτερα το Συμβούλιο και δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα ως προς την, ε, το επαγγελματικό δελτίο. Αυτή τη στιγμή μπορεί να συνταχθεί επαγγελματικό δελτίο, η λεγόμενη επαγγελματική κάρτα για τη συνεχή κατάρτιση. Τα κράτη-μέλη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να υπάρχει αυτόματη αναργό, αναγνώριση, με για το κοινό πλαίσιο κατάρτισης το οποίο χρειάζεται για να ε, συνταχθεί η επαγγελματική κάρτα. Η κατεξιοδότηση πράξης προβλέπουν αυτή την κατάρτιση και το κοινό αυτό πλαίσιο ισχύει για την αυτόματη αναγνώριση αυτό το ζητήσαν οι επαγγελματικοί κύκλοι, ιδιαίτερα για τη μαθητεία, για τα στάζ. Ιδιαίτερα αν ε, γίνονται σε τρίτο κράτος. Δηλαδή να υπάρχει αναγνώριση και σύμβαση για τις κατεξιοδότηση πράξεις για την αυτόματη αναγνώριση προσόντων κάναμε μία εξαίρεση για τις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές, γιατί ξέρετε ότι αυτό, αυτός ο φάκελος είναι δύσκολος. Αντίθετα, είχαμε ενίσχυση όλων των διατάξεων για τον, για τον νέο κατάλογο αρμοδιοτήτων των νοσηλευτών. Και η παρούσα οδηγία προβλέπει ότι οι τροποποίησεις αυτές δεν έχουν επιπτώσει στο νομοθετικό πλαίσιο των κρατών. Μέσα στα πλαίσια των προσαρμογών ίσονης, ίσονος σημασίας. Ως προς τους επαγγελματικούς κλάδους ήρθα σε επαφή με τους αρμόδιους και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω διότι κατά τους ε, μακρύς μήνες διαπραγματεύσαν. Είχαμε διαβουλεύσεις και προχωρήσαμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παρόντες. Νομίζω ότι κάναμε ένα μεγάλο βήμα για την επαγγελματική κινητικότητα, για τις υπηρεσίες και για να χτίσουμε την εμπιστοσύνη για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Ε, το αυθόρμητο χειροκρότημα δείχνει την εκτίμηση όλων. Ο Κρίστιαν Μπουζόη αποχώρησε από το Κοινοβούλιο, διότι είναι πρόεδρος στη Ρουμανία της ε, ε, Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας. Θα ήθελα να εγκρίνετε το πακέτο ηλεκτρονικά και έτσι θα ελέγξουμε και το σύστημά μας για να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουμε υπεράριθμους. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία για να εγκρίνουμε το συνολικό πακέτο για την οδηγία των επαγγελματικών προσόντων. Έχουμε 41 παρόντες, 42 ε, σοσιαλιστές ένας υπεράριθμος, κάποιος να αποσύρθει και είναι κάποιος που έχει εισαγάγει την κάρτα του αλλά δεν ψηφίζει. Ποιος είναι αυτός ή δεν ε, λειτουργεί το μηχάνημά σας. that was rather strange. Did somebody decide not to vote? The NI won over. εγγεγραμμένοι έχουν έναν υπεράριθμο, παρακαλώ να αποσυρθεί. Ε, ε, right, so 39. 39 σύνολο. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 37 υπέρ και 2 αποχές. Σας ευχαριστώ. Αυτή η επίσημη συμφωνία θα προωθηθεί στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Τέλος, σε αυτό το τομέα, σε αυτό το, στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, θέλαμε να σας το υποβάλουμε σήμερα, αλλά αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη έχουν μπλοκάρει γιατί έχουμε να κάνουμε με κατεξουσιοδότηση πράξης και εκτελεστικές πράξεις. ήμουν σε, ήρθα σε επαφή με τον κύριο Λένε που ήρθε σε επαφή με τον Επίτροπο Σεύκοβιτς. Μίλος, μίλησα με τη Γενική Διεύθυνση και ελπίζουμε να επανέλθουμε το Σεπτέμβρη. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να προωθήσουμε το θέμα. Αν θέλετε λεπτομέρειες θα τα πούμε μετά διμερός. Ωραία. Ψηφοφορίες λοιπόν. πρόταση για πρόταση Γκέπχαρτ και Χανς Πέτερ Μάιερ δύσκολη ε, θα είναι αυτή η ψηφοφορία ξέρω ότι οι εισηγητές και η γραμματεία εργάστηκαν θα ήθελα να εργάστηκαν σκληρά, θα ήθελα να γίνει μια ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δεν ξέρω κατά πόσο οι θέλουν το λόγο, αλλιώ περνάμε στις ψηφοφορίε. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Η πρώτη είναι να απορρίψουμε την πρόταση της Επιτροπής. Αρχίζει η ψηφοφορία για την ε, τροπολογία 339, για απόρριψη. 40 κάρτες. Απορρίπτεται. Τώρα προχωράμε στην άλλη, στην επόμενη ψηφοφορία ηλεκτρονικά και πάλι θέμα αρχής γιατί θα δούμε ποια μπλοκ θα μας απασχολήσουν. Να αλλάξουμε τον κανονισμό σε οδηγία. Τροπολογία 16 Gephardt. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 41 τώρα. Πέρας και εγκρίνεται 22 υπέρ 17 κατά. Άρα προχωρούμε για το μπλοκ Α, στο μπλοκ Α, προφορική 1 Hans Peter Mayer. Ποιοι είναι υπέρ. Ας το κάνουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία υπαριθμών 1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρία εξήντα τρία. υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Άρα οι δύο καταπίπτει. Τρία υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 4, 5 και 6 on block υπέρ, κατά, εγκρίνονται. 64 δεν την ψηφίζουμε, 65 υπέρ. 65. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 65. Σας παρακαλώ να ψηφίσετε πιο γρήγορα. Σοσιαλιστές ένας υπεράριθμος. Πέρας. Εγκρίνεται 21 έναντι 27. Εάν ψηφίσετε, θα ήθελα να ψηφίσετε αμέσως γιατί χάνουμε χρόνο. Και εάν ε, οι κάρτες δεν χρησιμοποιούνται, να τις βγάλετε παρακαλώ. 61 Γκέπχαρτ αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Ωραία. Εγκρίνεται 67 Gephardt. Αρχίζει η ψηφοφορία. Βλέπω ότι προχωρούμε με την ταχύτητα του φωτός. Έξοχα. Εγκρίνεται. 68 καταπίπτει 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 71 του κυρίου Μάιερ υπέρ. Αρχίζει η ψηφοφορία, με συγχωρείτε, ηλεκτρονικά θα το δούμε. Πέρας. Απορρίπτεται 8 των εισηγητών υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 72 και 73 δεν τις ψηφίζουμε. Τροπολογία 2 των δύο εισηγητών. Αρχίζει ψηφοφορία για την 2. Πέρας. Απορρίπτεται. 76. Αρχίζει ψηφοφορία για την 76. Πέρας. Απορρίπτεται. Επίσης, 77 και 84 τα Πάμε στην 85. 85. Όχι, 87. Λέει ο πρόεδρος το ελέγχο γιατί δεν ξέρω. 86. Or we just vote on They are together. Right. 86 and 87 are together. Sorry. So 86, 86 and 87. 86 και 87 για συντακτικές αλλαγές. 85. Άρχεται η ψηφοφορία για την 85. Πέρας. Απορρίπτεται. 9. Ε, ναι, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 370 αρχίζει η ψηφοφορία για την 370 πέρας απορρίπτεται 88 Αρχίζει η ψηφοφορία για την 88. Θα ήθελα να επιταχύνετε κάπως απορρίπτεται. 88, 90, 89 και 90 ε, εγκρίνονται αυτόματα. 13 υπέρ κατά εγκρίνεται. 371 αρχίζει η ψηφοφορία για την 371. Πέρας απορρίπτεται. Έχουμε πολλές διαγραφές και φτάνουμε στην 100. Hans Peter Mayer αρχίζει η ψηφοφορία για την 100. Πέρας. Απορρίπτεται. 101 μέχρι 109 διαγραφές 388 το. Α, με συγχωρείτε, 109. 109, με συγχωρείτε. 109. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 109. Εγκρίνεται. Άρα έχουμε μία σειρά διαγραφών και φτάνουμε στην 388. 388. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 388 ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται με άνεση. 389 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Στο παράρτημα 1 έχουμε μία σειρά διαγραφών. Άρα φτάμε στην προφορική 3. 4, 4. Προφορική 4. Αρχίζει η ψηφοφορία για την προφορική 4. Πέρας ε, καταπίπτει. Γιατί έχουμε ισοψηφία. Έχουμε μία σειρά διαγραφών στη συνέχεια. Άρα πάμε στην 452. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 452. Πέρας. Εγκρίνεται. 173. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 174. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται. 176. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. 179. Υπέρ. Σας παρακαλώ, σηκώστε τα χέρια σας να δω. Όχι, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Με ανάταση χειρό. Γιατί έχουμε πολλές ομάδες. Και με πολλές διαφορετικές απόψεις. Τότε να ψηφίζουμε λίγο πιο γρήγορα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, Πρόεδρε. Να κάνετε, να κάνετε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 453 του κυρίου Κρόιτσμαν έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 454 του κυρίου Βάινχολτσερ. Υπέρ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 455 του κυρίου Κρότσμαν. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 180 του κύριου Μάιερ. Η ψηφοφορία καλό. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 181. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 183. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 182 ως προσθήκη. Ως προσθήκη. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 185. Ψηφίζουμε. Πέρας, εγκρίνεται. 456 ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 184 καταπίπτει, 186 δεν ψηφίσατε, 187 λοιπόν. 184 ως προσθήκη, α, συγγνώμη. Μάλιστα, υπέρ. Όχι, ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Την 184 παρακαλώ ηλεκτρονικά ως προσθήκη, γρήγορα. Πέρας. Απορρίπτεται. 186-187. Α, συγγνώμη, είχε εγκριθεί 186-187. Ένα ψηφορία, παρακαλώ. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 188-189, λοιπόν. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. εγκρίνεται. 190. Ο 193. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 193. Πέρας. Εγκρίνεται. 194. 194 παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με σαφήνεια. Η 460 καταπίπτει, 195 υπέρ. Με τα χέρια, με τα χέρια. Διάνοτα ισχυρός. 195 υπέρ. Α ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Αν ο κύριος Μάντερ κάνει σαφέ ε, σήμα, θα καταλαβαίνω πιο καλύτερα. Ε, μάλιστα, απορρίπτεται με τρει ψήφου. Η 14. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 196. Υπέρ. Όχι, όχι. Ηλεκτρονικά. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να ψηφίζουμε νομίζω με τις κάρτες. Σας παρακαλώ να ψηφίζουμε λίγο πιο γρήγορα. Πέρας ψηφοφορίας Τέσσερα 461. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Φτάσαμε και σε μία συμβιβαστική. Υπέρ. Όχι, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ γιατί είναι συμβαστική 1. Εγκρίνεται. Η 462 καταπίπτει λοιπόν. Και... Περνάμε τώρα στην 203, λέει ο πρόεδρος. Όχι. Στη 203. Στη 203. 204-205 από κοινού. Έναρξη ψηφοφορία. 203-204-205. Ηλεκτρονικά. Πέρα. Εγκρίνονται. 464. Υπέρ. Κατά. Τι κάνουν οι φιλελεύθεροι. Α, μάλιστα. Απορρίπτεται. 206. Υπέρ. Τι κάνουν παρακαλώ οι φιλελεύθεροι. Α, μάλιστα. Έχουμε εδώ πέρα πρόβλημα με δύο φιλελεύθερους. Πού έχουμε φτάσει τώρα. Αφαιρέθηκα. 206. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τη 206. Σας παρακαλώ λίγο πιο γρήγορα. Πέρας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται 206. 207 δεν ψηφίζουμε. 208. Εγκρίνεται αυτόματα η 207. Άρα τι κάνουμε, την ψηφίζουμε την 208. Όχι. 209 λοιπόν έπεσε αυτό. Η 210 λοιπόν. Η 210. Να ψηφίσουμε λοιπόν 210. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 211. Την ψηφίζουμε. Έναρξη ψηφορίας. Πέρα. Και αυτή εγκρίνεται. Η 212, 213. 213. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρα. Εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε τη συμβαστική B3. Hans Peter Mayer. Α, μάλιστα, πίπτη, γιατί εγκρίθηκε η 213. Και έτσι περνάμε στην 200, στην 469. 469. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. 216, 217, 218 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. 15. Τι 15 να ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 219, 220, 221. Όχι, δεν τις ψηφίζουμε αυτές. Αυτομάτως συγκρίνονται. 222 ε, λοιπόν τώρα. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέρα. Εγκρίνεται. 223. Υπέρ. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Νομίζω ότι δεν έχουμε περιθώριο, πρέπει να ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Είναι δύσκολε οι ισορροπίε και αλλάζουν και συνέχεια. Για την 223 λοιπόν. Έναρξη ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. 224, όχι συγγνώμη, 225. Του κυρίου Μάιερ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται με σαφήνεια. 472. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 470. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 471. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 473. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 226. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 474, 475, 476, 477 και ούτω καθεξής. Καταπίπτουν όλες. Και περνάμε στην 227. 227 υπέρ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Καταπέπτει και τη 227. Πάμε στην 235-236. Α, μάλιστα. So we can vote on them. So we need to vote on 228 πρέπει να ψηφίσουμε την 229 ξεχωριστά. Α, συγγνώμη, την 228 και την 229 από κοινού. Με παρακολουθείτε, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 230, 232, 235, 236 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 237 και το καθεξής, μάλιστα ναι, πίπτου Πάμε στην 257, υπέρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 488 του κυρίου Ρόσπο. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 489 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2,64 υπέρ. Σας παρακαλώ σηκώνετε καλά τα χέρια κατά. Εγκρίνεται. Άλλο ένα μεγάλο μπλοκ. Μέχρι το 2,72 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Έλεγχος. Να το ελέγξουμε. Οκ. Okay για την 272 παρακαλώ έναρξη ηλεκτρονική ψηφορία. Απορρίπτεται. 273 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 274 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 275 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 277 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 278 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 279 Καταπίστη. 280. Να ψηφίσουμε και την 282. Μόνο το δεύτερο τμήμα. Παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 283. 493. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 288 τώρα. Υπέρ. Α, η 286, συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Την 286 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε τον 288, την 288 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 289 καταπίπτει, 290 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 494 ή 293 τώρα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 496 καταπίτσι και η 294 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301. Πάμε στην 498 αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Συμφωνείτε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι προτάσεις σα, Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Και τώρα από προσμιουργικές σκέψη. 17 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Κατά. Μάλιστα, εγκρίνεται με σαφή διαφορά. Δεν μπορούμε να τους ψηφίσουμε από μαζί, μπορούμε. Οι επόμενε δύο ναι. Οι 18 και 19 λοιπόν μαζί. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 3.40, 3.41, 3.42 του κ. Ροσφόρ. Από κοινού. Παρακαλώ υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 20, 21. 21, 23 μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 47-3-48 από κοινού παρακαλώ υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Πολλέ διαγραφέ διαγραφές έχουμε Διαγραφέ διαγραφέ. διαγραφές. 5. 375-378 από κοινού παρακαλώ. 357-358 παρακαλώ. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Τώρα λοιπόν ψηφίζουμε το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότησης ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 22 ψήφοι υπέρ, 17 κατά, μία αποχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, να πάρουμε το λόγο μήπω οι εισηγητέ πριν περάσουμε στην επόμενη ψηφοφορία. Κάποιος από του δύο εισηγητέ θέλει το λόγο μήπω. Η κυρία Γκέπχαρτ. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συνεργάτες, τους ε, συναδέλφου για την καλή συνεργασία και τον Hans Peter Mayer παρά το γεγονό ότι επί του προηγουμένου ήταν πραγματικά εκ διαμέτρων διαφορετικές οι απόψει μας καταφέραμε να συνεργαστούμε με τη μέθοδο τη συνέντευξη παρά το γεγονό ότι δεν ψηφίσαμε από εκείνο. Νομίζω ότι είναι καλό να συμβαίνουν έτσι τα πράγματα και πιστεύω ότι η ψηφοφορία που μόλι ολοκληρώσαμε ε, πέτυχε δύο βασικούς, πολύ βασικούς στόχους. Με τις πολλές διαγραφές που κάναμε, καταφέραμε αυτά που με την οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή τα είχαμε δημιουργήσει και αυτά που είχαμε πετύχει με την έκθεση SWAP να μην τα θέσουμε υπό αμφισβήτηση και να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο η προστασία του καταναλωτή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και κατά δεύτερον, να μην προκύψει ένα προαιρετικό σύστημα, να μην προκύψει νομική αβεβαιότητα, να μην έχει ο καταναλωτής ε, την ανασφάλεια του να βρίσκεται σε μια ασαφή κατάσταση και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας είχαν επισημάνει ότι αυτό θα συνέφερε. Και νομίζω λοιπόν ότι η Επιτροπή μας έδρασε υπέρ του συμφέροντος ε, των καταναλωτών και ψήφισε προς την κατεύθυνση αυτή. Και τώρα φυσικά καλώ και τους συναδέλφους από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων να κάτσουν να σκεφτούν επίσης πώς θα συνεχίσουν τη διαδικασία αυτή, πώς θα θέλουν να τοποθετηθούν για το θέμα αυτό είναι σαφή η τοποθέτηση νομίζω, πολύ πιο σαφής από ό,τι περίμενα να την σεβαστούν λοιπόν την τοποθέτησή μας αυτή και να συμπεριλάβουν την γνωμοδότησή μας στη δική του απόφαση. Ιδάλω θα το πούμε στην Ολομέλεια, δεν υπάρχει άλλη λύση. Ευχαριστώ. Και ίσω να προσθέσω ένα τελευταίο στοιχείο, αν μου επιτρέπετε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, βοηθούς και όλους τους υπαλλήλους. Είχαμε εδώ δύο φακέλους ενωμένους σε έναν. Δεν ήταν καθόλου απλή η επεξεργασία τους. Να ευχαριστήσω πραγματικά τους υπαλλήλους της Επιτροπής, οι οποίοι έκαναν εξαιρετική δουλειά. Ήταν πραγματικά δύσκολο το έργο και μας βοήθησαν ιδιαίτερος. Αλλά και τους υπαλλήλου της ομάδας μου και του δικού μου, του γραφείου. Γιατί ακόμα και η προετοιμασία του καταλόγου ψηφοφορίας ήταν πραγματικά πολύ περίπλοκο έργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Μάιερ, ήταν σαφές εξ αρχής ότι ήταν δύο διαφορετικές ε, ε, διαμέτρου οι απόψει μας και γι' αυτό λοιπόν ε, το θέμα ήταν θα πάμε προς το α ή προς το β. και όσοι ήταν φυσικά υπέρ του Α δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν το Β. Και το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν ε, αρκετά σαφές. Κρίμα που έχασε η ενιαία αγορά. Γιατί ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να κάνουμε με τον νόμο αυτό ήταν να ανοίξουμε την αγορά. Να παρέχουμε πιο μεγάλη προσφορά στον καταναλωτή. Δεν το πετύχαμε αυτό. Και δεν νομίζω ότι το αποτέλεσμα επί του περιεχομένου το οποίο ψηφίστηκε πρόκειται να γίνει αποδεκτό από το Συμβούλιο. Γιατί το προσπαθήσαμε άλλωστε και πριν από δύο χρόνια. Το Συμβούλιο δεν το αποδέχτηκε. Δεν νομίζω ότι μετά από δύο χρόνια θα έχει αλλάξει εκ βάθρων η τοποθέτηση του Συμβουλίου. Έχω την εντύπωση ότι κάτι ψηφίσαμε εμεί πολύ ωραίο, ενίσχυση του εθνικού δικαίου προστασίας του καταναλωτή και στη τελική ανάλυση δεν βγάλαμε τίποτα. Θα το δούμε, θα το δούμε αυτό πάρα πολύ σύντομα και νομίζω ότι θα φανεί μέσα στην τρέχουσα θετία. Κάτι άλλο τώρα. Ψηφίσαμε πολλά πράγματα για τα οποία δεν είμαστε αρμόδιοι λόγω αποκλειστικότητας. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να τα ψηφίσουμε. Αν ψηφίσει διαφορετικά η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, το θέμα είναι αγαπητή Εβελίν. λέτε να λάβει υπόψη η Γιούρη, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, ε, τη δική μας γνωμοδίτηση. Η Επιτροπή Γιούρη ασφαλώ θα μας πει, κοιτάξτε, εμείς είμαστε αποκλειστικά αρμόδιοι. Ούτε εκεί λοιπόν θα είναι αρκετά σαφές τι θα γίνει. Κρίμα, κρίμα. Εδώ είμαστε υπεύθυνοι και αρμόδιοι και για την προστασία του καταναλωτή αλλά και για την ενιαία αγορά. Και τώρα επιλέξαμε την προστασία του καταναλωτή σε εθνικό επίπεδο, όχι την εσωτερική αγορά. Κρίμα. Είχαμε πριν από κάποια χρόνια ένα μεγάλο όραμα για την διεύρυνση και την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς. Λοιπόν, αυτό το όραμα το υπονομεύσαμε σήμερα. Κρίμα. Λυπάμαι. Να σας το πω ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει όραμα για τις συνοριακές δραστηριότητες. Αυτό το αφήσαμε. Α, ψηφίσαμε μόνο αλλαγή του εσωτερικού, εθνικού δικαίου ήταν πολύ στενή η θεώρηση του θέματος και δεν μπορούμε με τον τρόπο αυτό να διαμορφώσουμε την Ευρώπη. Είμαι απόλυτα πεπισμένος γι' αυτό. Αλλά εννοείται ότι σεβόμαστε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εδώ στην Επιτροπή και πραγματικά ανυπομονώ να δω τι θα γίνει στις υπόλοιπες Επιτροπές και στο Συμβούλιο. Good. Well, as, um, as you out, this is... Όπως είπατε, είναι μια γνωμοδότηση στην Επιτροπή Νομικών. Αύριο από τις 9.30 μέχρι τη 1 υπάρχει εργαστήριο με τα Εθνικά Κοινοβούλια για πρόταση ε, κοινού ευρωπαϊκού δικαίου πολίσεων. Ο κύριος Μπερλιγκέρ θα μιλήσει. Δεν ξέρω αν η κυρία Γκέπχαρτ ε, μπορεί να μας, να μας δώσει τη δυνατότητα να εκφράσουμε και εμείς τη δική μας άποψη. Εγώ θα ήθελα να είμαι εκεί για να πω την άποψη μου. κύριο Σφαμπ, Από ό,τι κατάλαβα, ο συνάδελφος προηγουμένως ε, τάχθηκε υπέρ της πρότασης, όχι? Αυτό είναι ο τίτλος του σεμιναρίου που σας ανέφερα προηγουμένως. Μπορεί με τη σημερινή ψηφοφορία να τους δείχνουμε ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος και ίσως άμα το ήξεραν στην Επιτροπή των νομικών υποθέσεων μπορεί να το παρουσιάσουν ε, κατά αυτή την έννοια ε, και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Τέλος πάντων. 4Q1. Αύριο στις 9.30. Με μία. Αν θέλει κανείς λεπτομέρειες, δεν ξέρω αν η κυρία Γκέπχαρτ έχει προσκληθεί ή όχι. Ε, όχι, λέει η κυρία Γκέπχαρτ, αλλά θα πάω. Και ο κύριος Μάιερ θα είναι εκεί. Περνάμε τώρα σε μία ακόμη σημαντική έκθεση πρωτοβουλίας για τα επόμενα βήματα της εσωτερικής αγοράς. Ε, οι συγκητές έκαναν μεγάλη προσπάθεια για τις μοιβαστικές τροπολογίες. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε γενικές γραμμές νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή η ατμόσφαιρα, πολλέ συμβαστικέ τροπολογίε, Κάποιοι μάλιστα απέσυραν κάποια σημεία τα οποία θεωρούσαν ε, ότι έπρεπε να αλλάξουν, ε, γιατί εγώ ήθελα μερικά σημεία να τα διατηρήσω ισχυρά, να στείλω ισχυρά μηνύματα στα κράτη-μέλη. Δεν είναι δυνατόν να στερούμε, να, στερούμαστε, να στερούμε από τους ε, Ευρωπαίους πολίτες θέσεις απασχόλησης και γι' αυτό θα ήθελα να έχω μια πραγματικά ανοιχτή αγορά υπηρεσιών στην Ευρώπη. Να ευχαριστήσω την Πύργη, τον Θιερή από το ΕΛΚ και τη Γραμματεία και όλους τους υπόλοιπους βοηθούς ε, που με βοήθησαν πάρα πολύ να φτάσω στους συμβιβασμούς και να έχω ένα κείμενο το οποίο είναι ισχυρό και σαφές. Μία προφορική τροπολογία θα έχουμε για τη συμβιβαστική 15. Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποσύρατε την 59. Θα το διαβάσω όταν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, αλλά να ευχαριστήσω και εσάς για την κατανόησή σας. Περιμένουμε αγωνία την ψηφοφορία. Ωραία. Λοιπόν, συμβαστική 4, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 29 Χόλτσερ, Να ελέγξουμε ηλεκτρονικώς. Έναρξη ψηφοφορίας. 41 τώρα ψηφίζουν. Το ΕΛΚ έχει έναν ε, υπεράριθμο. Ωραία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30, πουπάκι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 4 της Επιτροπής ΕΜΠΛΕ. Είναι συμβατή, είναι συμβατή. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 34. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 35. Έχει αποσυρθεί. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 19. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται 39 έχει αποσυρθεί. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην ε, τροπολογία 2 της Επιτροπής Απασχόλησης. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έμπλ 1 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. πλού 3 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. πλού 5 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 45, 46 έχουν αποσυρθεί. Α, όχι, 45 δεν έχει αποσυρθεί. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Τη 45 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Έμπλε 9 ναι, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έμπλε 6 7 υπέρ. Κατά. Ε, απορρίπτεται. Η 54 τώρα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 59 έχει αποσυρθεί. 60. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Employment 11. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 65. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικό στην 65. Ψηφίζουμε. Πέρασα. Απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 70 και 71 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 125. Σωστά. Με προφορική τροπολογία. Του ΕΛΚ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 77. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Employment 12. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 78. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 79 έχει μια προσθήκη υπέρ, κατά. 80 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Υπάρχει προφορική τροπολογία εδώ. Κυρία Κορατσαμπίλτ, ναι. Αφορά τη συμβαστική 15, διαβα... προσθέτω ενημερώνοντας ε, τους πολίτες ε, και τις επιχειρήσεις για τα δικαιώματά τους που προκύπτουν από την, ε, υπηρεσία, από την οδηγία υπηρεσιών. Συμφωνείτε όλοι? Ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Employment 14, λέει ο Πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 86. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 87 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 89. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Employment 8 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 10 employment υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 90-91 υπέρ κατά απορρίπτονται. 92 υπέρ κατά εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά εγκρίνεται με διαφορά. 98 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά εγκρίνεται. Πάμε στην 114 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 116 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 118 υπέρ κατά εγκρίνεται 119 υπέρ κατά απορρίπτεται 120 υπέρ κατά απορρίπτεται 121 υπέρ κατά εγκρίνεται 122 υπέρ κατά απορρίπτεται 123 έχει αποσυρθεί 124 ε, Υπέρ. Κατά. Πορύπτεται. 126. Με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 127. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 132. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη τολογικές σκέψεις. Συμβιβαστική 1. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Employment A και B έχουν καλυφθεί. τροπολογία 9 υπέρ κατά εγκρίνεται. Employment B υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά υπέρ 12 υπέρ υπέρ υπέρ υπέρ τις 12 να ψηφίσουμε ηλεκτρονικό στη 12. Έναξη ψηφοφορίας. Πέραση. Εγρίνεται 23-15. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά εγκρίνεται 20 υπέρ κατά εγκρίνεται. Λοιπόν, αιτιολογικές σκέψεις, όλες μαζί υπέρ κατά απορρίπτονται έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για το σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται 23 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και 13 αποχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Εύλην. Θα ήθελα να πω στην ομάδα μου ότι θεωρώ ότι είναι κρίμα Πολλές από τις συμβιβαστικές τροπολογίες ή τι τροπολογίες που είχαν υποβληθεί για κοινωνική προστασία, που είναι σημαντικές για την εσωτερική αγορά, δυστυχώ καταψηφίστηκαν. Εγώ θα το θέσω και πάλι αυτό στην Ολομέλεια και ελπίζω ότι σε συνεργασία με άλλες ομάδες μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εκδοχή του κειμένου. Κύριε Κορατσαμπίλ, στη συγγήτρια. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με τη... Ε, ε, χαίρομαι πολύ με τη συνεργασία που είχαμε την κυρία Ράπτη και με την κυρία ε, Γκέμπχαρτ. Δούλεψαν πολύ για την έκθεση αυτή. Αυτή τη στιγμή αποφασίσαμε επί συμβιβαστικών τροπολογιών, τις οποίες λάβαμε υπόψη όλες τις ανησυχίες. Κάθε συμβιβαστική τροπολογία από τις 18 εγκρίθηκε από τους σοσιαλιστές. Όταν βλέπω ότι υπάρχουν 13 εποχές ε, από τους σοσιαλιστές, αναρωτιέμαι πόσο αξιόπιστο είναι το κείμενο και πόσο μπορούμε στο μέλλον ε, να εμπιστευόμαστε το γεγονός ότι όταν καταλήγουμε σε μια συμφωνία γίνεται σεβαστή. Με εξέπληξε αυτό, ελπίζω να συνεχίσουμε με καλό πνεύμα συνεργασίας ε, και ανοιχτό πνεύμα Μάλιστα εγγράφως οι σοσιαλιστές ε, με ευχαρίστησαν για την ευελιξία και την κατανόησή μου. 13 αποχέ για μένα, ε, τι να πω, ε, για μένα χρήζει εξηγήσεων αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ακούσατε ήδη την εξήγηση. Επειδή θα ψηφίσουμε και στην Ολομέλεια, είναι μια ε, έκθεση πρωτοβουλίας, ε, οπότε αν έχουμε συνένεση πριν από την Ολομέλεια θα είναι καλά. Κυρία Γκέπχαρτ. Δεν μπορώ να δεχθώ αυτό το παράπονο της κυρίας Κοράτσα Βίλτ. 18 συμβαστικές τροπολογίες, ναι, τις εγκρίναμε όλες, συμφωνήσαμε, συνεργαστήκαμε για αυτές, αλλά υπήρχαν αρκετοί τομείς που έχουν να κάνουν με την κοινωνική προστασία για τις οποίες ε, η δική σας ε, ομάδα δεν πρόσφερε κανένα συμβιβασμό. Χάσαμε όλες αυτές τις ψηφοφορίες και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι είναι τα πράγματα στην πολιτική ζωή. Τι να κάνουμε τώρα. Θα υποβάλουμε τροπολογίες για την Ολομέλεια για τους τομείς αυτούς και ελπίζω να υπάρξει συμβιβαστική λύση μαζί με την ομάδα σας. Μέχρι τότε. Ελπίζω να τα καταφέρουμε, λέει ο Πρόεδρος. Κοιτάξτε, δεν θέλω να ανοίξουμε συζήτηση τώρα για αυτό το θέμα. Ε, ο καθένα έχει πει την άποψή του. Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο θέμα τώρα. Έχουμε να ψηφίσουμε την έκθεση του κυρίου Μάντερς για την απλοποίηση της μεταφοράς μηχανοκίνητων οχημάτων ταξινομημένων σε άλλο κράτος μέλος εντός της ενιαίας αγοράς. θέλετε να πάρετε το λόγο, κύριε Μάντερς. από ό,τι κατάλαβα, αν περάσει τροπολογία 23, έχετε μια πρόταση για μελέτη αντικτύπου, αν κατάλαβα καλά, έτσι. Ωραία, σας δώσω το λόγο τότε. Λοιπόν, πρώτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 59. Κατά. Υπέρ. Υπέρ πρώτα. Υπέρ πρώτα. Α, συμφωνείτε. Μάλιστα. Τροπολογία 59 υπέρ, επαναλαμβάνω. Κάτω. Υπέρ πάλι. Υπέρ Τις 59 επαναλαμβάνει ο πρόεδρος. Κατά. Εγκρίνεται. 60. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 9. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 62 καταπίπτει. 10 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 63-64 καταπίπτουν 11. Υπέρ. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικός. Την 11. Πέρα στις ψηφοφορίες. 36 υπέρ. Συγγνώμη, αλλάξτε γνώμη. Ε, πού να το ξέρω. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Γκρίνεται. 13 υπέρ κατά εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά απορρίπτεται. 66 καταπίπτει. Συμβαστική 25 υπέρ κατά εγκρίνεται. 10 ε, ε, συμβαστική υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Transport 9 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ, κατά εγκρίνεται, συμβιβαστική 12 υπέρ κατά εγκρίνεται, 16, 17 ε, μαζί υπέρ κατά εγκρίνονται, transport 10 κατά πίπτη, 18 υπέρ κατά εγκρίνεται, 19 κατά πίπτη, 11 υπέρ κατά εγκρίνεται, συμβαστική 14 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τη συμβιβαστική 15, 23 και 16 μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί. Α, καλά, τη 15 μόνη της τότε. Συμβιβαστική μόνη της, 15. Υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ναι, κύριε Σιγητά. θέλουμε να θέσουμε ως όρο οι συντονιστές σήμερα να δεχθούν ε, μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων για αυτό το θέμα. Εάν αυτό εγκριθεί λοιπόν, λέει ο Πρόεδρος, ε, θα κάνετε μία πρόταση ε, μελέτης αντικτύπου στους συντονιστές. Λοιπόν, 23, συμβαστική. υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Α. 86 καταπίπτει. 18 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τρανσπορτ 15 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 94 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 35. Η 94 απορρίφθηκε. Στη 35 είμαστε τώρα. Ψηφίζουμε 35 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 36 και 37 μαζί. Όχι. Καλά. 36 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, 43. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 24. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 46. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τράνσπορτ 22 καταπίπτει, 47 καταπίπτει, 48. 48 ψηφίζουμε, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 26 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τρανσπορτ 23. 24, συγγνώμη, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τρανσπορτ 25 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 110 καταπίπτει. Πάμε τώρα στα παραρτήματα. 50. Υπέρ. Κατά. Τι θέλετε, να τις πάρουμε όλες μαζί, να τις ψηφίσουμε. Μπορούμε να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες του παραρτήματος μαζί, των παραρτημάτων. Λοιπόν, όλες μαζί. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αιτιολογικές αναφορές. 52, υπέρ. 52 υπέρ. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 18-18. Τρεις δεν ψήφισαν. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Γκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 και 2. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί. Ναι. Ωραία. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Η συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Transport 5 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 5. Ωραία, συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 πίπτη. Συμβιβαστική τροπολογία 8 και 6 μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί. 8 και 6 λέει έχουν ψηφιστεί, έχουν εγκριθεί, συγγνώμη. Now, eight is, eight according to us is automatically. Η 8 εγκρίνεται αυτομάτως γιατί η 20 εγκρίθηκε με την τροπολογία 38, άρα πρέπει να ψηφίσουμε τη συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικώς το σύνολο της έκθεσης. Τρεις κάρτες είναι εντός των μηχανημάτων χωρίς να έχουν ψηφίσει συνάδελφοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. 34 ψήφοι υπέρ, ε, κανένας, καμία ψήφος κατά και τρεις αποχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή. Α, ο κύριος Α, ο Μάντες, ο κύριος Μάντες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες ε, που υποστήριξαν με ευρύτατη πλειοψηφία και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αρχίσουν οι άτυπες διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή και το Συμβούλιο γιατί θέλουν να αρχίσουν ήδη τις διαπραγματεύσεις και βρισκόμαστε πολύ μπροστά έναντι του Συμβουλίου. Νομίζω ότι αυτό είναι θέμα συντονιστών που θα συζητήσετε απόψε. Εάν θέλετε λοιπόν μπορείτε να προσέλθετε στους συντονιστές για να υποβάλλετε την ε, πρότασή σας στους συντονιστές και θα ψηφιστεί το Σεπτέμβριο. Οι συντονιστές ε, το δέχονται. Δεν έχει νόημα να ε, επισπεύσουμε αποφάσεις σήμερα. Πρόταση για τη στρατηγική ασφάλεια του χωρου ένας ανοιχτός, ασφαλής και προστατευόμενος ε, κυβερνοχώρος. Ο κύριος Σφάπ είναι εισηγητής και θα ήθελα να λάβει το λόγο πριν ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους και τις συναδέλφους που συνεργάστηκαν για τις προτάσεις συμβιβασμού. Ευχαριστώ την ε, γραμματεία και τους ε, συνεργάτες. Από την ε, τελευταία εβδομάδα ίσως δεν διαβάσαν όλοι το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. εν πάση περιπτώσει έχουν προβληθεί πολλές αιτιολογήσεις των συμβιβασμών. Με τις προφορικές δεν έχω πρόβλημα. Καταρχήν, εάν όμως τις δεχτώ, τότε οι συμβασμοί δεν θα λάβουν πλειοψηφία. Γι' αυτό δεν είμαι και ιδιαίτερα ενθουσιώδης για τη συμπερίληψή τους. Μίλησα και με τον συνάδελφο Ραμόν και πιστεύω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε, να προβάλλουμε ξεχωριστή ψηφοφορία. Εάν δηλαδή ενταχθούν στους συμβιβασμούς θα πρέπει να αντιταχθώ. Ζητώ, συγγνώμη, λυπούμε γι' αυτό, αλλά ίσως στην Ολομέλεια όλοι ταχθούν υπέρ. για να καταλάβω τι λέμε για τις προφορικές. Εσείς λέτε ότι αντιτάσσεστε, δεν θέλετε καν να ψηφίσουν. Μπορούν να ψηφιστούν χωριστά. Αυτή είναι νέα απόφαση της Ολομέλειας, από ό,τι φαίνεται. So apparently Άρα δεν μπορούμε να τις ψηφίσουμε χωριστά. Έτσι έχει αποφανθεί η Ολομέλεια. Άρα το θέμα λύγει εδώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω τι συνέβη και πώς το θέμα σχετίζεται με τις σημερινές ψηφοφορίες. Εγώ έλαβα γνώση των ε, τροπολογιών συμβιβασμού που προτάθηκαν από τον κύριο Σβάμπ ε, την προηγούμενη Παρασκευή μόλις. Και χτες ε, μελέτησα τις τροπολογίες και πρότεινα ως ενιαία διαδικασία Ε, ε, την συμπερίληψη των προφορικών. Καταλαβαίνω τη θέση του κυρίου Σουβάμπ. Ίσως όμως ε, σε αυτή τη διαδικασία υπήρξε μεγάλη σπουδή. Δηλαδή υπήρξε σπουδή στον κυβερνοχώρο. και αυτό οδήγησε σε ένα τελικό διφορούμενο, ιδιαίτερα όσον αφορά ορισμένες τροπολογίες που είναι ύψης της σημασίας. Υπ' αυτή την έννοια, οι προφορικές που υποβλήθηκαν σε αυτή την Επιτροπή θα πρέπει να υποβληθούν ως πλήρης τροπολογία στην Ολομέλεια και έτσι ελπίζω να μην υπάρξει πρόβλημα. Μπορούμε να τις μεταφέρουμε στην ε, Ολομέλεια, διότι έχουν μεγάλη σημασία. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Θα ήθελα λοιπόν να τις λάβουμε υπόψη στην τελική ψηφοφορία. για να διασαφηνίσουμε την όλη διαδικασία Έτσι εργάζεται η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες για την Ολομέλεια. Άρα η πρόταση ψηφίσματος αν εγκριθεί θα πάει στην Ολομέλεια. δύο μέλη θα πρέπει να αντιταχθούν στις προφορικές. Άρα ο κύριος Σβάμπ δεν θέλει να ψηφιστούν οι, τρο... οι προφορικές, δηλαδή να ενταχθούν στο γενικότερο πλαίσιο. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες. Στις προφορικές θα δω κατά πόσο η Επιτροπή συμφωνεί. Υπάρχουν αρκετά μέλη προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε ταχύ ρυθμό, εν πάση περιπτώσει. Καταρχήν μια τεχνική υφής τροπολογία. Μπροκ και Κέλλαν που συνυπογράφουν τον, το ψήφισμα. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό. Στα στέχοντας υπόψη μπορούμε να τις δούμε όλες on block. Δηλαδή άφετ συν όλες όσες προέρχονται από αυτή την ε, Επιτροπή υπέρ κατά εγκρίνονται. Στέχοντας υπόψη 8 υπέρ κατά εγκρίνεται 10 υπέρ Νομίζω ότι θα πρέπει να ελέγξουμε. Τροπολογία 10. Ελέγχουμε. Μπορούμε να επιταχύνουμε παρακαλώ. Υπεράριθμοι από το ΕΛΚ. Εγκρίνεται 20 έναντι 15 και μία αποχή 12 υπέρ. Κατά εγκρίνεται στη συνέχεια προφορική της Επιτροπής Εξωτερικών ε, Υποθέσεων Β. Ποιοι είναι υπέρ, εγκρίνεται και μετά το Γ της ΑΦΕΤ υπέρ, κατά εγκρίνεται. Συμβασμός 1 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 20 και 21 υπέρ, κατά, κατά παρακαλώ, απορρίπτονται. 23 υπέρ, Ας ε, ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 23. Παρακαλώ βγάλτε την κάρτα σας αν δεν ψηφίζετε. Απορρίπτεται. 17-19. 22 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 24-25 αφέτ αμπλοκ υπέρ. Κατά εγκρίνονται. 30 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 29 ως προσθήκη υπέρ. Κατά εγκρίνονται. εγκρίνεται. Και καταπίπτει 28. Σύμβασμος 2 υπέρ κατά εγκρίνεται 31 υπέρ κατά Σύμβασμος 3 υπέρ κατά εγκρίνεται 4 με ξεχωριστή που ζήτησαν οι φιλελεύθεροι. Ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα της 4 υπέρ κατά εγκρίνεται τμήμα 2 υπέρ, υπέρ, κατά, επίσης εγκρίνεται. 35, α όχι κατά καταπίπτει, συμβασμός 5 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά Υπέρ παρακαλώ του συμβασμού 6 κατά. Σαφώς εγκρίνεται. 44 υπέρ. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 44 αρχίζει η ψηφοφορία. 19 υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται. σε 7 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 53 με ξεχωριστή ψηφοφορία. Τμήμα 1 υπέρ, κατά. Σας παρακαλώ χέρια, υπέρ, κατά Απορρίπτεται σαφώς. Τμήμα δεύτερο υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Άρα 55 είναι προσθήκη υπέρ. Κατά Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε. 55. Απορρίπτεται. 61. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται σαφώς. Συμβασμός 8 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. 68 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 69 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά κατά τώρα κατά παρακαλώ ψηφίσατε δύο φορές μερικοί υπέρ Σίμψον τώρα κατά πάλι απορρίπτεται 72 υπέρ. Είναι διαφορετική σειρά χεριών. Αρχίζουμε λοιπόν, ελέγχουμε ηλεκτρονικά, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. 72. Πέρας. Απορρίφθηκε. 17 έναντι 19 και μία αποχή. 74 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 75 υπέρ κατά απορρίπτεται 76 α δεν ψηφίσω όχι 75 απορρίφθηκε άρα η 76 δεν μπορεί να θεωρηθεί προσθήκη όχι, όχι, είναι μόνη της ε, υπέρ κατά εγκρίνεται 77 υπέρ κατά εγκρίνεται 78 ως προσθήκη υπέρ. Κατά εγκρίνεται 79 ως προσθήκη υπέρ. Κατά εγκρίνεται 80 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 81. ένα. Άφετ πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ εγκρίνεται 81 υπέρ κατά νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά πρέπει να ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας ε, η ισοψηφία απορρίπτεται 82 υπέρ κατά απορρίπτεται σαφώς 84 υπέρ απορρίπτεται 83 υπέρ υπέρ κοντά είμαστε ψηφίζουμε για την 83 ελέγχουμε ηλεκτρονικά πέρας περνάει με μία, με μία ψήφο διαφορά 86 υπέρ κατά εγκρίνεται 89 υπέρ κατά απορρίπτεται 87 υπέρ κατά απορρίπτεται 88 υπέρ κατά εγκρίνεται 90 υπέρ κατά απορρίπτεται 91 υπέρ κατά Απορρίπτεται. Απορρίφθηκε, ναι, ναι. 95 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 93 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 94 ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται. 97 υπέρ εγκρίνεται. 96-98 υπέρ κατά εγκρίνονται. Συμβασμό 9 υπέρ εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά απορρίπτεται. 102 υπέρ κατά απορρίπτεται. 103 υπέρ κατά εγκρίνεται. Αφέτε παράγραφος 20 για διαγραφή υπέρ. Hm. Ας ελέγξουμε, ας ελέγξουμε. 21. Αφέτε διαγραφή. Ας δούμε. Πέρας. Απορρίπτεται για μία ψήφο. 104 υπέρ. 104 ας ελέγξουμε. pp 1 over. Ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ, ένας υπεράριθμος. Βγάλτε την κάρτα σας αν δεν ψηφίζετε. απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 107 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε καλύτερα. 107 ελέγχουμε. Ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ. Ε, απορρίπτεται για δύο ψήφους. 108 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 109 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 110 ως προσθήκη υπέρ, κατά εγκρίνεται. 111 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Συμβασμός 10 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβασμός 11 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 120 υπέρ. Κατά. Νομίζω πρέπει να ελέγξουμε. 120 ελέγχουμε. Πέρας απορρίπτεται για δύο ψήφους, ε, συμβιβασμός 12, ξεχωριστή ψηφοφορία, τμήμα 1, υπέρ, κατά, εγκρίνεται, τμήμα 2, υπέρ, κατά, νομίζω ότι εγκρίθηκε. 123 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 124 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 125 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 127-28 υπέρ. Κατά αποχές. Πώς ψηφίζει το ΕΛΚ. 127-128 υπέρ κατά εγκρίνονται. 129 υπέρ. Νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 129. Πού πήγατε, πού πήγαν όλοι, φεύγουν. 33, 34, πέρας, εγκρίνεται. Άρα ψηφίζουμε το σύνολο της πρότασης ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται με 33 ψήφους υπέρ 2 κατά και μία αποχή. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σβάπ. Θα δούμε τι θα γίνει με τις τροπο, τροπολογίες στην Ολομέλεια. Έκθεση Γκαλό. Στη συνέχεια ε, λυπάμαι που γίνεται αυτή η σύμπτυξη. Θα το δούμε το συντομότερο δυνατόν. Ε, κυρία Γκαλό, θέλετε κάτι να μας πείτε για την έκθεση η συγγήτρια παρακαλώ για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά. Όχι κύριε Πρόεδρε, δεν έχω τίποτα ιδιαίτερο να πω. Απλώς να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις που συνεργάστηκαν επί του θέματος. Σας ευχαριστώ. Ωραία, αρχίζουμε. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 75. Καταπίπτει 74 προσθετική υπέρ. Κατά. Α, όχι καταπίπτει. 76. Υπέρ. Κατά. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρέπτεται, αλλά θα το ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 76. Σας παρακαλώ λίγο πιο γρήγορα, γιατί δεν θα προλάβουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 7 ως προσθέκη υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 83 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 84 καταπίπτει. 85 υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κα, Κατά. Εγκρίνεται. 88 καταπίπτει λοιπόν. Η 11 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 89 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 12 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 90 και η Γιούρια 17 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η Λίμπε 14 καταπίπτει, η 91 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 93 υπέρ. Η 93. Νομίζω θα χρειαστεί να ψηφίσουμε χρονικά. Γιατί 93 θα είναι οριακό το αποτέλεσμα. Είστε, παρακαλώ γρήγορα. 33 ψηφίζουν. Πέρα ψηφορίας. Απορρίπτεται με διαφορά δύο ψήφων. Την 92 τώρα να ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Λίμπε 15. Ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 94 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 13 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 95 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η γύρω 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 97 διαγραφή υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας το ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά παρακαλώ ψηφίζουμε. 33 ψηφίζουν, απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 99 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. παρακαλώ. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 99. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Γιούρι 22 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 108. Υπέρ. Κατά. Α. Εγκρίνεται. 109. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 110. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Σεμιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 113 του κυρίου Κρόιτσμαν. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 114 υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. Η 20 της κυρίας Γκάλο υπέρ. Κατά. Αχάθηκα μισό λεπτό λέει ο πρόεδρος. Στην 20 της κυρίας Γκάλο. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 115 καταπίπτει. 116 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 117. Με την ψηφίζουμε 21. Της κυρίας Γκάλο υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 118 και 119 συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 23 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι επόμενες 3. Η 124. Α, συγγνώμη, η 100. 122, Mr. του κυρίου Κρότσμαν ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 124. Υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 24 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 126 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 130 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 131. Καταπίπτει 132 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 133 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 134 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 135 υπέρ, κατά, έγκρινεται. 137 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 138 υπέρ, κατά, υπέρ, κατά, το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Για την 138. Δεν ήταν σαφέ το αποτέλεσμα. Πέρα ψηφοφορία. Έχουμε λοιπόν, ε, εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. 26 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 27 και 139 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 140 και 141 καταπίπτουν. Συμβιβαστική 8. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Η 29 το κυρία Γκάλο υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Η 30 και 146 υπέρ. Κατά εγκρίνονται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Η 151 καταπίπτει. Η 32. Η 32. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 152. Καταπίτη. Ως προσθήκη. Αναφέρεται στην άλλη σελίδα. Η 152 ως προσθήκη, κυρία Πεντρικάστη, μάλιστα. Η 152 ως προσθήκη, λοιπόν, ψηφίζουμε υπέρ κατά εγκρίνεται διαφορά. Η 153 καταπληκτή. Η 153 υπέρ κατά απορρίπτεται. 154 155 υπέρ κατά εγκρίνεται. 156 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Δεν είναι σαφέ τι κάνουν οι ελληνικέ ομάδε. Για την 162 παρακαλώ ηλεκτρονικά να ψηφίσουμε. Πέρα. Απορρίπτεται. 163 υπέρ κατά το ίδιο είναι το αποτέλεσμα απορρίπτεται 164 τώρα υπέρ κατά απορρίπτεται επίση. 165 του κυρίου Κρότσμαν υπέρ κατά απορρίπτεται η 34 της κυρίας Γκάλο υπέρ δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Κατά λάθος ψηφίσαμε την 165 γιατί αυτόματα απορρίπτεται η 167 του κ. Κρόιτσμαν υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 34 της κυρίας Γκάλο υπέρ. Κατά. Και αυτή εγκρίνεται. 169 της κυρίας Γκάλο. Και 170 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 171-172 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 173 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 175 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται 176 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται 177 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Adopted, that's oh, right. Εγκρίνεται, συγγνώμη. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Η 178 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 179 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 180 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 181 και 182 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 183 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα για την 183 υπέρ. Υπέρ. Ψηφίζει το ECR. Κατά δεν είναι καθόλου σαφές. Δεν είδα να σηκώνει κανείς από πίσω τα χέρια. Να ψηφίσουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 183 πρώτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με τη λέξη significant, υπέρ του significant, κατά, εγκρίνεται. 184 υπέρ κατά εγκρίνεται 185 υπέρ κατά απορρίπτεται 186 υπέρ κατά εγκρίνεται 187 υπέρ κατά απορρίπτεται 188 υπέρ κατά εγκρίνεται 189 υπέρ κατά εγκρίνεται 190 υπέρ κατά εγκρίνεται 193 υπέρ κατά απορρίπτεται 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 ως προσθήκη ως προσθήκη 192 υπέρ κατά απορρίπτεται σε τμήματα την 195 πρώτο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται και αν έχουμε διαφωνία. Μάλλον το in case of some national doubt, το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 197 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 196 ως προσθήκη υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Η 198 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Η 199 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 200 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 215 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 216 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 40 και 217 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 41 υπέρ κατά εγκρίνεται 219 υπέρ κατά εγκρίνεται 220 υπέρ κατά απορρίπτεται 221 222-223 23, μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί, θεωρείτε. 2, 21, 22, 23, υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 2.24. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2.25 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2.26 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2.28. 29 συγγνώμη υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Να ψηφίσουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 229. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 231. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Η 230. Η 230. Υπέρ. Για τη 230 παρακαλώ, είσαστε υπέρ, κατά, δεν είναι σαφές. Εγκρίνεται. Η 232. Η 232 λέει ο πρόεδρος υπέρ, κατά εγκρίνεται. Η 235 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Η 238 του κυρίου Σβάμπ. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 241 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η συμβαστική 12 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Λείπε 50. Ως προστίκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 45 και η 51 υπέρ κατά εγκρίνονται. 46, 245, 72, 52, υπέρ. Κατά εγκρίνονται. 246 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 248 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Για την 248 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Κατά. Απορρίπτεται, συγγνώμη. Η 249 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Γύρω 17. 73, συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 250 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 254 υπέρ. Α, συγγνώμη, 252. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 254 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 253 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 255 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 256 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 257 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 258 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 261 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 262 με προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ. Κα... Υπέρ παρακαλώ. Υπέρ, υπέρ. Κατά. Έγκρινεται. 263, 264 καταπίπτουν, 267 υπέρ. Κατά. Έγκρινεται. 266 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 47 και η λίμπε 53 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 268 ως προσθήκη υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 269. καταπιπτει Η 270 καταπίπτει. falls if 268 is adopted. 268 was adopted. But no, is 270. 268 was adopted. It has a consequence on 269 and 270, which both fall. All right, okay. So according to us, 270 falls. Καταπίπτει η 270 μου λένε. 48 και λείπει 54 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 271 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 49 και το καθεξής. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και όλοι οι υπόλοιποι. λιπε 56. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 274 ως προσθήκη υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 276 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Η 277 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 280 με προφορική τροπολογία υπέρ, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 282 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 292 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 293 καταπίπτει, 294 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Η 297 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 298 με προφορική τροπολογία υπέρ. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Η 299 ως προσθήκη υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Η 300 υπέρ. Α, η 50, η 50, συγγνώμη. Ψηφίζουμε την 50, υπέρ. Κατά. Έγκρινεται. Η 300, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 301, υπέρ. Κατά. Έγκρινεται. Η 302 και η 303, υπέρ. Υπέρ. Κατά. θα πρέπει να τις ελέγξουμε ενωριακό το αποτέλεσμα. Για την 302 και την 303 παρακαλώ. Απορρίπτονται. 304 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 51 και 52 τεχνικές ε, τροπολογίες. Η 53. 55, συγγνώμη. 55 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην 307 υπέρ Υπέρ για την 307 παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. Και περνάμε στα παραθύματα. Λίμπη 58 υπέρ. Κατά. Έγκρινεται. 308 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 309 υπέρ. Κατά. Κατά. Παρακαλώ. Οριακό, οριακό το αποτέλεσμα. Να ψηφίσουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά για την 309. Πέρασε. Απορρίπτεται. Λείπει 59 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 310 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 311 εγκρίνεται αυτόματα. Και περνάμε σε τελογικές σκέψεις λοιπόν. 56 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 57 λοιπόν καταπίπτει και οι υπόλοιπε καταπίπτουν. Περνάμε στην 58 ω προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 59 υπέρ. Κατά. Απορρίφεται. Η 60 υπέρ. Κατά. Ε, εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 62 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 64 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 63 ως προσθήκη παρακαλώ υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε τις επόμενες μαζί αν θέλετε. Μέχρι την 68 μέχρι και την 68, 65, 3, 66, 4, 5, 67, 68 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται όλες. 69 καταπίπτει, 70 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 71 υπέρ. Να ψηφίσουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Είναι δύσκολο, δύσκολη η ψηφοφορία για την τροπολογία του κ. Πέρας. 18 υπέρ 16 κατά. Εγκρίνεται. 72 και 73 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα λοιπόν θα ψηφίσουμε το σχέδιο της γνωμοδότησης στο σύνολό του. Ηλεκτρονικά. Ξεκινάμε την ψηφοφορία για την γνωμοδότηση της κυρίας Γκάλο για την Επιτροπή Βιομηχανίας. Μήπως κάποιος δεν έχει ψηφίσει. Ψήφισατε όλοι. Πέρα ψηφορίας. 31 ψήφοι υπέρ. Καμία ψήφος κατά και δύο αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Γκάλο. So, thank you very much indeed. ευχαριστούμε λοιπόν. Έχουμε δύο θέματα ακόμα στην διαδικασία διάταξή μας, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, αποχωρήστε ήσυχω. γιατί η κυρία Βάιλερ περιμένει να ξεκινήσει. Please, if you could let us get on with the next business, because we, we Αργήσαμε με τις ψηφοφορίες, οπότε να πάμε γρήγορα στα επόμενα θέματα. Συνήθως θέλω να είμαι στην ώρα μου, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερα σήμερα. Ζητώ συγγνώμη, ήταν περίπλοκες οι ψηφοφορίες. Έχουμε λοιπόν ε, μια σημαντική συζήτηση για τις τροπολογίες κυρίας Βάιλερ που είναι εδώ. Ο κύριος Φαντενκάμπ είναι εδώ. Ο κύριος Μάντερς είναι εδώ, η κυρία Ριούλα είναι εδώ, εγώ είμαι δύο, οπότε όλοι οι σκιώδεις είναι εδώ. Και βλέπω ότι και ο κύριος Ζηράου είναι εδώ. Κύριε Αρίας, μήπως μπορείτε να πάτε πιο εκεί γιατί δεν βλέπω. Λοιπόν, για να ακούσουμε από την κυρία Βάιλερ, ποια είναι η άποψή της για τις τροπολογίες. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλό θα ήταν να είχαν γίνει και άλλες ψηφοφορίες, γιατί θεωρώ ότι πριν το θερινό διάλειμμα συζητάμε ήδη τις τροπολογίες. Δεν μοιάζομαστε ιδιαίτερως, γιατί θα αποφασίσουμε μόλις τα τέλη Σεπτεμβρίου αλλά οι τροπολογίε θα πρέπει να εξεταστούν σε κάθε περίπτωση. Πέρα από την έκθεση έχουμε και 36 τροπολογίε και όλοι φροντίσαμε, νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι το φρόντισαν αυτό, να έχουμε μια συνένεση, αν θέλετε, και να συμφωνούμε, να συνάδουμε με το πακέτο Ρόιτοβα για το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Προκειμένου να υπάρχει ένα συντονισμός. Πέντε μικρά σημεία έχω να αναφέρω. Το πρώτο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η 116, τραπολογία 116. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης να σας πω ότι διαπίστωσα ότι για το θέμα αυτό, για το, το πρόβλημα αυτό, δεν υπάρχουν διαβλέψεις για την προστασία των καταναλωτών όπως για άλλα θέματα στην Γερμανία. Είναι υπεύθυνη και αρμόδια η υπηρεσία δικτύων. Αλλά δεν αισθάνονται πραγματικά αρμόδια και το ίδιο ισχύει και σε άλλες χώρες. Και γι' αυτό λοιπόν στην 116 συστήνουμε στα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν όχι μία υπηρεσία, αλλά να ορίσουν μία από τις υφιστάμενες υπηρεσίες ως αρμόδια. Να ορίσουν δηλαδή ε, μια υπηρεσία στην οποία μπορεί να απευθύνεται το καταναλωτή όταν έχει προβλήματα. Ή αν θέλει να α, δηλώσει κάποια προϊόντα κατά δεύτερον. Ένα δεύτερο θέμα που προέκυψε από τη συζήτηση με του κοιότητε συζητητέ ήταν το εξή. Ότι τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν διαφορετικές πραγματικότητες και διαφορετικά δεδομένα. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι ήταν ε, αποδεκτό να εξαιρεθεί ε, από το πεδίο εφαρμογή ε, με το θέμα της εκπομπής των υπηρεσιών εκπομπής μέχρι ότου κατάλαβα ότι στην Γαλλία για, και στην ε, Ισπανία για παράδειγμα διαφέρει κατάσταση από ότι στην Γερμανία και στην Ολλανδία όπου κάλυπτονται 100% γι' αυτό λοιπόν συμφωνήσαμε με την κυρία Φαντεγκάμπε να αποσυρθεί η τροπολογία 120 αλλά να διατηρηθεί εκ 16. Και αυτό βρίσκει σύμφωνους όλους μέσα στην Επιτροπή αλλά ικανοποιεί και όλες τις, επιτροπ... τις εταιρείε που επηρεάζονται. Το θέμα της ε, καταχώρησης νομίζω δεν υποστηρίζει, κανένα δεν υποστηρίζει κανένας από τους κοιόδης. Ξέρω ότι στο Συμβούλιο διαφέρει η κατάσταση και η μισή είναι υπέρ, η μισή είναι κατά, αλλά νομίζω ότι συνεπάγεται τόσο μεγάλο άχθος γραφειοκρατικό και κόστους που θεωρώ ότι πραγματικά είναι πραγματικά δυσανάλογο. Γι' αυτό και το αφαίρεσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ήθελε αυτό και κάποια κράτη-μέλη είναι υπέρ. Θα δούμε τι θα προκύψει από τις περαιτέρω διαβουλεύσεις, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι δεν βοηθάει στην παρούσα φάση. Τώρα, το επόμενο θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω Όχι, νομίζω ότι τελείωσα με τις τροπολογίες και με τις προτάσεις μου. Αυτά ήταν. Γενικά, κοιτάξτε, συμφωνούμε. Συμφωνούμε και μεταξύ των σκιωδών, γενικότερα, ότι θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα σε ό,τι αφορά τις συσκευές. Ξέρω ότι θα προτιμούσα να μην συμπεριληφθεί στην έκθεση αυτή, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα μήνυμα. Δεν είναι δυνατόν η παροχή πίσω από την πλάτη του Κοινοβουλίου να αποσύρουν συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε ό,τι αφορά αυτές τις ε, πρόσθετες συσκευές να κάνουν να βγάζουν μεγάλα κέρδη στην πλάτη του καταναλωτή γιατί γενικά υπάρχει μεγάλη συμφωνία μεταξύ των καταναλωτών ότι θα πρέπει να προκύψουν ε, επιτέλους να υπάρξουν ε, ενιαίες ομοιόμορφες συσκευές για τη φόρτιση των συσκευών. Νομίζω όμως ότι επί του συνόλου υπάρχει μια γενικότερη συνένεση. Ότι θέλουμε να αποστείλουμε το μήνυμα αυτό. Και βλέπω ότι στις τροπολογίες ότι σε γενικές γραμμές Συμφωνούμε. Και για αυτό το λόγο ακριβώς αλλάξαμε λίγο το χρονοδιάγραμμα με τους κοιόδησίτες. Στις 25 Σεπτεμβρίου θα γίνει εδώ στην Επιτροπή η επόμενη συζήτηση με συμβιβαστικές τροπολογίες και μπορούμε πολύ απλά αρχές Σεπτεμβρίου οι σκιώδεις ε, μαζί με τη Λιθουανική Προεδρία να κάτσουμε να συζητήσουμε αυτά και να τα υποβάλουμε και να τα συζητήσουμε στις 25 και νομίζω ότι μπορούμε άνετα να ψηφίσουμε στις 26 Σεπτεμβρίου. Ίσως θα καταφέρναμε να ολοκληρώσουμε και την ψηφοφορία στην Ολομέλεια μέσα στο τρέχον έτος, γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην το πετύχουμε. Όσο πιο νωρίς τα ολοκληρώσουμε αυτά, τόσο το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ για τις τροπολογίες και την παρουσίασή τους. Ε, ο κύριος Βαντεκάν πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Βάιλερ και να τη συγχαρώ για την ε, πολύ γερή ηγεσία της σε ό,τι αφορά αυτό το τεχνικό θέμα. Νομίζω ότι πραγματικά θα καταφέρουμε πάρα πολύ καλά. Κατά δεύτερον, Τη συγχαίρω για το πολύ φιλόδοξο χρονοδιάγραμμά τη. Πραγματικά θα ήταν εκπληκτικό αν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό με στο 2013. Κατά τρίτον, έχω και εγώ καταθέσει κάποιε τροπολογίε, κυρίω σε ό,τι αφορά το γραφειοκρατικό άχθο και τη μείωση αυτού. Και ανυπομονώ να δω πώς θα διαμορφωθούν οι συμβιβαστικές τροπολογίες και κατά πόσο θα διτηρηθεί αυτή η πρόθεσή μου στις συμβιβαστικές τροπολογίες. Στην παρούσα φάση δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Νομίζω ότι καλή είναι η δουλειά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομο να ευχαριστήσω την κυρία Βάιλερ για την πολύ καλή προσέγγιση της. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή στην έκθεση αυτή η αποστολή ενός μηνύματος σαφούς, όπως σας είπα, για την εναρμόνιση των συσκευών φόρτισης. Το ζητήσαμε ήδη στο παρελθόν ως Επιτροπή και υπάρχει και ένα μνημόνιο συνεννόησης. Θέλουμε λοιπόν να το προωθήσουμε. Η Nokia και η Apple δυστυχώ ε, δεν θέλουν να συμφωνήσουν και ζητούν επιπλέον κόστος. Κρίμα, κρίμα νομίζω ότι αυτό θα έπιθε πολύ τους πολίτες. Θέλω λοιπόν και χαίρομαι που συμπεριλαμβάνεται εκ νέου το θέμα αυτό και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να το προωθήσει. Είμαι πολύ ικανοποιημένος και ανυπομονώ να περάσουμε στην ψηφοφορία. Mrs. Ρούλα. Ναι. Δεν θέλει να πάρει το λόγο η κυρία Ρούλε. Λοιπόν, Είμαι και εγώ σκιώδης συζητητή, Να πω και εγώ ορισμένα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμότατη υποδοχή που επιφυλάξατε στι τροπολογίες μου. Ε, σκοπό είχαν να βελτιώσουν τι διαδικασίε και ιδιαίτερα να επιτρέπουν σε νέο εξοπλισμό να εμφανίζει όλες τις πληροφορίες ε, στην οθόνη του ίδιου του εξοπλισμού που νομίζω ότι μπορούν πολύ εύκολα να το κάνουν πολύ εξοπλισμοί, εξοπλισμοί σήμερα και είναι πολύ πιο εύκολο να διαβάζει κανεί ε, αυτέ τι πληροφορίε, στον εξοπλισμό στην οθόνη του εξοπλισμού. Αν δεν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο, α, βλέπω η κυρία Ρόιτοβα είναι εδώ, γιατί Έχουμε υπόψη μας και το νέο, τις, τις, πτυχές, τις νέες πτυχές, των, τις νέες νομοθετικές πτυχές του θέμα αυτού. Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει ορισμένα πράγματα για το πώς βλέπει την κατάσταση του πακέτου αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να κάνω ορισμένα σχόλια για τις νέες τροπολογίες. Ε, όσον αφορά την έκθεση, Παρουσιάσαμε ήδη τα ε, σχόλιά μας σε σχέση τώρα με τις νέες τροπολογίες. Συμφωνούμε σε γενικές γραμμές ε, οι περισσότερες, οι περισσότερες ε, τροπολογίες μας βρίσκουν σύμφωνους. Τέσσερα, τέσσερα σημεία θα ήθελα να θέσω μόνο. Πρώτον, σε σχέση με την τροπολογία 118, από ό,τι καταλάβαμε η τροπολογία 120 αποσύρθηκε. Υπάρχει όμως ακόμη μια τροπολογία που αφορά τον, ε, την εξαίρεση των, ε, ε, των θορύβων των ακουστικών. Αυτό μας φαίνεται λίγο προβληματικό, γιατί η απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου ήταν ένας από τους στόχους μας. Η εφαρμογή της οδηγίας ε, ήταν δυσχερής γιατί κάποια ακουστικά ήταν εντός, κάποια ακουστικά ήταν εκτός. Ο στόχος ήταν αυτή η οδηγία να αφορούσε μόνο τους ε, ε, μεταδότες, αλλά τώρα λέμε να αναφέρονται μόνο τα ακουστικά. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά πρέπει να συμπεριλάβουμε όλα τα ακουστικά στην οδηγία. και αν πρέπει να δούμε τις ε, παραμέτρους, ε, ας τις δούμε εντός του ιδίου νομοθετικού ε, κειμένου και να μην υπάρχει διαφορά μεταξύ της, του ραδιοεξοπλισμού και ε, των, της οδηγίας EMC, γιατί είχε δημιουργήσει προβλήματα για την, τις, τους φορείς εποπτείας της αγοράς και στους κατασκευαστές. Όσον αφορά τώρα τους φορτιστές κινητών τηλεφώνων. Κοιτάξτε, προτείνεται μεταξύ των βασικών ε, απαιτήσεων που υπάρχουν ήδη. Είναι το άρθρο 3 παράγραφος 3α. Οι βασικές απαιτήσεις είναι η διαλειτουργικότητα. Έχουμε μία εκτίμηση επιπτώσεων ε, για να δούμε κατά πόσο Ε, τα tablets και ε, οι φορητοί υπολογιστές, τι θέση πρέπει να έχουν και να δούμε τις ε, διάφορες δυνατές πρωτοβουλίες. Γιατί ξέρετε ότι το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, όλες οι δυνατότητες είναι στη διάθεσή μας και θελοντικές συμφωνίες όσο εκκρεμούν τα αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα της κατάστασης στις αρχές του επόμενου έτους. Αν θέλετε όμως να επιμείνετε σε συγκεκριμένα στοιχεία ε, σε συγκεκριμένα είδη ραδιοεξοπλισμού, εμείς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είναι στι βασικέ απαιτήσει, αλλά στα παρατήματα, γιατί οι βασικές απαιτήσει καλύπτουν τα πάντα. Σε σχέση τώρα με την τροπολογία που λέει ότι κάθε αδιοεξοπλισμός ε, πρέπει να έχει και έναν οικουμενικής χρήσης φορτιστή. Αν γίνεται κάτι τέτοιο, δεν χρειάζεται να, το αναφέρουμε, να το συνδέουμε με κάθε είδος ραδιοεξοπλισμού για λόγους περιβαλλοντικούς. Άμα έχουμε έναν φορτιστή μπορούμε να το χρησιμοποιούμε για όλα. Μία ακόμη προβληματική τροπολογία είναι 99. Lex Specialis. Είναι μια τομεακή οδηγία αυτή και η τροπολογία αυτή για μας δικαιολογείται σε οριζόντιο νομοθετικό κείμενο. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο, τότε το πιο συγκεκριμένο ισχύει. Αλλά αυτό είναι ήδη τομεακή οδηγία, οπότε μας φαίνεται ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε σχέση με την υπόλοιπη τομεακή νομοθεσία. Τι είναι το ειδικό τώρα, ο εξοπλισμός ή η άλλη τομεακή οδηγία σε σχέση τώρα με την ηλεκτρονική σήμανση. Το καταλαβαίνουμε αυτό και αναφερόμαστε στις τροπολογίες 103 και 111 το έχουμε συζητήσει πολλές φορές ε, με τους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων φορέων και τους εκπροσώπους των κρατών μελών. Ε, υπάρχουν πρακτικά προβλήματα που δεν έχουν ακόμη επιληθεί σε σχέση με αυτό. Και το πρακτικό πρόβλημα είναι ότι οι καταναλωτές και οι αρχές εποπτείας αγοράς ε, θέλουν να βλέπουν την πληροφορία πριν αγοράσουν το προϊόν αυτά που έχουμε για την ηλεκτρονική σήμανση είναι ότι πρέπει να λειτουργήσει κανείς το προϊόν για να μπορεί να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες. Σε σχέση, για παράδειγμα, με κάποια από τα προϊόντα που έχουν ε, μπαταρία, που δουλεύουν με μπαταρία. Πρέπει κάποιος να φορτίσει πρώτα την μπαταρία για να μπορέσει να ελέγξει μετά την πληροφορία, τις πληροφορίες. Και αυτό είναι το πρακτικό πρόβλημα που δεν μπορούμε ακόμη να επιλύσουμε ε, ούτε και οι κατασκευαστές μας μπορούν να το επιλύσουν αυτό. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα στην πρακτικότητα αυτή τη λύση για την ηλεκτρονική αγορά για την ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαρίστω ε, να σα διαθέσουμε ε, άλλα έγγραφα ή να ε, δώσουμε περαιτέρω διευκρινήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, θετική σας προσέγγιση. Βέβαια, απογοητεύομαι κάπως που η τροπολογία μου ε, θεωρείται ότι είναι πολύ προηγμένη για την τωρινή τεχνολογία. Κρίμα, αλλά ίσως να μπορέσουμε να σας πείσουμε κάποια στιγμή, να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση όπως κάναμε και σε άλλες περιπτώσεις στη συνεργασία μας μαζί σας. Αν δεν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο, να δώσω το λόγο στην κυρία Βάιλερ να συνοψίσει και μετά ε, να μας πει οτιδήποτε άλλο θέλει. Επειδή συμφωνούμε όλοι για τα θέματα αυτά, να σας πω ότι βρισκόμαστε σε φάση επικοδομητικών συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξετάζουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφορών διατάξεων, εξετάζουμε τι ε, είναι χρήσιμο, τι θα ωφελούσε του καταναλωτέ. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια φάση πολύ επικοδομητικού διαλόγου και γιατί το τονίζω αυτό, γιατί έχω μια τελευταία παρατήρηση να κάνω. Δεν έχουν μείνει πολλοί συνάδελφοι, αλλά είναι οι αρμόδιοι εδώ και είναι και ο πρόεδρο τη Επιτροπή να σα πω ότι είμαι στο Κοινοβούλιο εδώ και πολύ, πολλά χρόνια. Αλλά για πρώτη φορά έμαθα εδώ πέρα στο θέμα αυτό κάτι το οποίο πραγματικά με εξέπληξε οι επιστολές, τα mail, τα τηλεφωνήματα των, υπηρεσιών, των εταιριών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι κάτι το οποίο όλοι το γνωρίζουμε, αλλά για πρώτη φορά, Πρόεδρε, έλαβα μία επιστολή όπου μου έγραψε ένας βιομηχανικός σύνδεσμος και μας είπε ότι δεν βρήκε εξετάζοντας τις τροπολογίες του ε, κειμένου του ψηφίσματος δεν βρήκε να αποτυπώνονται οι δικές της τροπολογίες. Πραγματικά έμεινα άφωνη. Αυτό τι αποδεικνύει, ότι κάποιοι βιομηχανικοί σύνδεσμοι πιστεύουν ότι αρκεί να μας γράψουν κάποιες προτάσεις για να τις μεριλάβουμε. Καλέ οι διαβουλεύσει, καλέ και ο επικοδομητικό διάλογο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς ως ε, βουλευτές ε, αυτόματα προασπίζουμε αυτά που μα προτείνουν. Πραγματικά έμεινα άναυδη. Τους ε, έγραψα ένα αντίστοιχο απαντητικό γράμμα, αλλά πραγματικά το τονίζω αυτό, γιατί πραγματικά πρώτη φορά σε 20 χρόνια μου συνέβη αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας επίστησατε την προσοχή σε αυτό. Υπήρξαν πολλές συζητήσεις σε σχέση με την ε, η ικανότητα των μελών της Επιτροπής να υποβάλουν ε, τοπολογίες αν πρέπει να την αντιγράφουν και να την επικολούν από άλλες πηγές, γιατί όταν πρόκειται και γνωμοδοτήσεις εμπειρογνώμων, προφανώς λαμβάνουμε υπόψη όλα αυτά που μας ε, στέλνουν ως ιδέες ε, εξωτερική της Επιτροπής μας. Πρέπει να αναθεωρήσουμε πολύ καλά τις τροπολογίες πριν τις υποβάλουμε και ελπίζω να γίνει αυτό. Αλλά ευχαριστούμε πολύ που μας το είπατε αυτό. Όπως είπε η κυρία Βάιλερ, ε, συμφωνήσαμε και μιλάω για το σκιώδης ηγητής ε, να προτάξουμε την έγκριση στις 26 Σεπτεμβρίου που θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με τη Λιθουανική Προεδρία και να προχωρήσουμε για αυτό το σημαντικό φάκελο. Γιατί πρέπει να υπάρξει συμφωνία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 We have your Ναι, υπάρχει ουγγρική καμπίνα από ό,τι φαίνεται. He's just, no, no, just waiting to get the go ahead for you. Περιμένουμε δύο λεπτά να λυθούν τα τεχνικά προβλήματα. Δύο λεπτά και μετά θα πάρετε το λόγο. Προσπαθούμε να λύσουμε τα περιδιαμηνία στις της κυρίας Καλπάτσου. Κύριος Μάντερς θέλει να πάρει το λόγο. Πολύ απλό είναι. Έχω κάποιες πληροφορίες ε, από Γερμανούς επιρρογνώμενες. Μου στείλαν αυτή την πινακίδα αυτοκινήτου. Αύριο έρχεται εδώ. Όποιοι θέλετε, 10 η ώρα, ε, θα μας δώσει σχετικές πληροφορίες. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Η κυρία Γκελπάτσο είναι η εισηγήτριά μας ε, για το θέμα του Γενικού Προπολογισμού. Η κυρία Ρούλε είναι εδώ. Εγώ βλέπω ότι μάλλον είμαι ο μόνος ε, σκιώδης εισηγητής εκτός από την κυρία Ρούλε. Να δώσω λοιπόν το λόγο στην εισηγήτρια να μας πει πώς πάνε τα πράγματα σε σχέση με τον προπολογισμό. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι για μένα είναι μεγάλη μου χαρά να σας παρουσιάσω το ψήφισμα για τον προπολογισμό του 2014. Όπως τα ξέρετε ασφαλώς, καλύψαμε μεγάλη απόσταση μέχρι ότου συλλέξουμε τα συγκεκριμένα δεδομένα, τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, γιατί μόλις ε, πριν από δύο εβδομάδες μας δημοσίευσε, μας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σχετικά στοιχεία. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την γραμματεία της Επιτροπής ε, ΙΜΚΟ, αλλά και τους υπαλλήλους από πλευράς του Λαϊκού Κόμματος, γιατί μας επέτρεψαν εξ αρχής να ορίσουμε τις βασικές προτεραιότητες και έτσι δεν χρειάστηκε να κινηθούμε στα τυφλά για μεγάλο διάστημα. Και έτσι λοιπόν καταφέραμε να ορίσουμε τα βασικά πολιτικά προγράμματα, τα, τα βασικά μέτρα, τα οποία είχαμε εξετάσει και στην προηγούμενη συνάντηση συνεδρίαση της Επιτροπής. Δεν θα μπω λοιπόν στα στοιχεία αυτά τα οποία έχουμε ήδη αναφέρει. Στόχος είναι να σας παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησης και να σας δώσω κάποια βασικά αριθμητικά στοιχεία. Οι συνάδελφοι έχουν μπροστά τους ε, τα βασικά αριθμητικά στοιχεία και νομίζω ότι καθίσταται σαφές ότι μόνο σε λίγα σημεία αντιμετωπίζουμε περικοπές. Αυτό είναι καλή βάση και σημείο αφετηρίας. Τέσσερις ε, σελίδες του σχεδίου προπολογισμού εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας, το δικό μας. Και εγώ θα πρέπει να προετοιμάσω μόνο μία πρόταση σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση για τα ιδρύματα πιστοποίησης και να σας πω γιατί ε, υπέβαλα τέτοια τροπολογία στην ε, Ευρώπη είναι μεγάλη η τεχνολογική εξέλιξη και σε όλο τον κόσμο βέβαια και γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντική η τυποποίηση προκειμένου λοιπόν να διασφαλίσουμε την σχετική ανάπτυξη προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προϊόντων, να διασφαλίσουμε την προστασία της υγείας των ε, πολιτών. Χρειαζόμαστε λοιπόν άλλα πρότυπα και ενιαία πρότυπα κυρίως σε όλη την Ευρώπη και φυσικά είναι πολύ σημαντικές οι επαφές ε, με, τα σχετικά, με τις σχετικές υπηρεσίες καθορισμού προτύπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το 20% που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρώ ότι δεν είναι αποδεκτό. Γι' αυτό λοιπόν υπέβαλα σχετική τροπολογία. Ξέρω ότι πρέπει ασφαλώς να δικαιολογήσουμε από πού θα βρούμε τους πόρους για το 20% αυτό που εκρεμεί. Βλέπω ότι στη γραμμή του προϋπολογισμού γίνεται, μάλλον επιτρέπεται μεταφορά των κονδυλίων. Σημαντική είναι ασφαλώς και η επένδυση στις ε, μικρομεσίες ε, επιχειρήσεις, αλλά οι δεσμεύσει είναι σπλαντικότερες από τις πληρωμές εδώ πέρα στην Επιτροπή και θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί να υπάρξει μια μεταφορά κονδυλίων στην γραμμή 12.010 βλέπω ότι Έχουμε τέτοια δυνατότητα μέσω της χρηματοδότησης του Solvit λοιπά. Και όταν περνάμε, αν περάσουμε ήδη στα μέσα, να σας αναφέρω κάτι το οποίο το κοιτάξαμε και στην προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής, το Europe Travel. Πρόκειται για μια ξεχωριστή παράγραφο και αυτό το πολιτικό πρόγραμμα μας ε, απασχόλησε ιδιαίτερως. Έγινε διαβουλεύσεις και προτάθηκαν κάποιες ε, τροπολογίες τις οποίες και μπορώ να αποδεχτώ. Παρακαλώ και τους συναδέλφους το ίδιο να πράξουν. Και όπως θα θυμούνται ασφαλώς οι συνάδελφοι, πρόκειται για ένα πολιτικό πρόγραμμα που προβλέπει ε, εφαρμογές για smartphones, εφή τηλέφωνα, για να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν οι πολίτε τέτοιες συσκευέ και στο εξωτερικό, στι διακοπέ του. Διατύφοντας τι τρει μεγάλε γλώσσε αυτέ αυτές οι τροπολογίες, αλλά και σε άλλε ευρωπαϊκέ γλώσσε. Και η σημασία των χρήσεων και των εφαρμογών στα κινητά τηλέφωνα, αλλά και των χρηστών τέτοιων εφαρμογών, αυξάνονται ραγδαία. πρόκειται για τομεί ε, που περιλαμβάνουν διάφορες, ε, μάλλον περισσότερα έτη χρηματοδοτικά. Έχουμε και το πρόγραμμα προστασία των καταναλωτών και διαπιστώνουμε ότι και στα δύο προγράμματα πρέπει να κάνουμε μειώσεις της τάξης του 5% σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μπορούμε φυσικά να χαρούμε με αυτό, αλλά εφόσον βρισκόμαστε σε εποχές περικοπών, δεχόμαστε την μείωση αυτή. Ένα μόνο σημείο θα ήθελα να αναφέρω ακόμα. Ένα πρόγραμμα online διατησία. πρόκειται για ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης με 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Να ευχαριστήσω τον ε, πρόεδρο Harbour για την επιστολή στην οποία διατύπωσε και έδειξε το θέμα αυτό. Και ο κύριος Επίτροπος ε, το έθεσε το θέμα αυτό γιατί το θεωρεί σημαντικό. Στην παρούσα φάση δεν γνωρίζουμε ακόμα πώς το ODR θα μπορέσει να συνεχίσει να χρηματοδοτείται. Όλοι φυσικά υποστηρίζουν τους τομείς που τους ενδιαφέρουν πιο πολύ. Δεν βλέπουμε να υπάρχει περιθώριο χρηματοδότησης από άλλους τομείς. Η χρηματοδότηση του ODR λοιπόν παραμένει ένα εκρεμές ζήτημα. Ίσως με την πάροδο του χρόνου ανακύψουν κάποιες λύσεις. Εγώ ανησυχώ γιατί δεν μπορώ ακόμα να βρω κάποιο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε το πρόγραμμα αυτό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία αυτή, αλλά πραγματικά πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο. Και άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη γνωμοδότηση. Γενικώ, πώς πρέπει να πω ότι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε νέες, ε, νέους κλάδους στην παιδιαρμοδιότητά μας και να μπορούν να χρηματοδοτείται αυτή οι κλάδοι. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βετερηθεί, αν μη τι άλλο, ο αρχικός φάκελος χρηματοδότησης. Και γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ τους συναδέλφους να με υποστηρίξουν προς την κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και θα χαρώ να ακούσω και τις δικές σας παρατηρήσεις των σκιωδών εισηγητών. Ευχαριστώ. Good. Well, Σας ευχαριστώ πολύ για την λεπτομερή σας εργασία η οποία βοήθησε ιδιαίτερα και ξέρω ότι υπάρχουν αμφιβολίες για τα τελικά ποσά που θα διατεθούν. Νομίζω όμως ότι έχουμε να κάνουμε με ένα βασικό σχέδιο όπου ήμασταν ιδιαίτερα αποδοτικοί και θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε τα πλαίσια μας. Λοιπόν, ο κύριος ε, Γκαρσία Ραμών έχει το λόγο. Ας αρχίσουμε με τους κοιόδης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ε, εισηγήτρια για την ε, παρουσίασή της προς την Επιτροπή καθώς και την πρόταση ψηφίσματος. Σε γενικές γραμμές ε, συμπίπτουμε, υπάρχει σύμπτωση απόψεων σε σχέση με τις προτεραιότητες που διαγράφονται και που είναι οι ίδιες και για μας. Θα ήθελα απλούστατα να ζητήσω τα αριθμητικά στοιχεία, πλήρη αριθμητικά στοιχεία και να προβάλλω και μία σκέψη σε σχέση με το σύνολο των δημοσιονομικών στοιχείων και του όγκου τους της Επιτροπής ε, ΙΝΚΟ από την αρχή της ε, θητείας μας, δηλαδή από το 2009 μέχρι το 2013 9 με 13 έτσι ώστε να ξέρουμε ποια ήταν η εξελικτική πορεία. Δηλαδή τα οικονομικά στοιχεία και η πρικοδότηση της ε, ΙΜΚΟ από τον ε, Γενικό Προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και στη συνέχεια να ε, γνωρίζουμε πώς είχε η εξελικτική πορεία, δηλαδή ποια ήταν η πρικοδότηση του ε, προϋπολογισμού με ορίζοντα το 2014 διότι προβάλλεται μείωση του συνολικού προϋπολογισμού της Επιτροπής ΙΜΚΟ. Αυτή είναι μια γενική πρώτη σκέψη. Δεύτερον, εγκρίναμε φέτος το 13 την ατζέντα των Ευρωπαίων καταναλωτών για την περίοδο 14-20. Θα ήθελα λοιπόν με περισσότερες λεπτομέρειες να δούμε πώς, ε, ποια ήταν η εξελικτική πορεία αυτής της ατζέντα και αν θα υπάρξουν ε, επιπτώσεις επί του προϋπολογισμού σε σχέση με τις προτάσεις επί τάπητος. και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να προβάλλουμε και τροποποίησεις. Ποιες είναι δηλαδή οι δυνατότητες που διαγράφονται. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι στο πιλωτικό σχέδιο σχέδιο σε σχέση με τα προπαρασκευαστικά μέτρα τα οποία προετοιμάζονται, θεωρώ ότι οι οργανισμοί πιστοποίησης θα πρέπει να δούμε κατά πόσο έχουν ε, πραγματική ε, πρικοδότηση και χρηματοδότηση όπως χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές ανάγκες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σμιτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια ασχολήθηκα με αυτό το θέμα γιατί ο Κριστιανό Μπουσόη εγκατέλειψε την ομάδα και το κοινοβούλιο υποστηρίζω τα πάντα και ιδιαίτερα τα τελευταία σχόλια, δηλαδή τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές όπως προδιαγράφονται, γιατί αυτό είναι ύψης της ε, σημασίας. Δεν με βρήκε σύμφωνο η απόφαση προηγούμενης εβδομάδας, αλλά νομίζω ότι θα βρούμε κάποια λύση το Σεπτέμβριο για τις ΜΜΕ βεβαίως. Ε, είχαμε μία ακρόαση με τον πρόεδρο Ντράγκη χτες και υπήρξαν μεγάλα ζητήματα για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Είπε ο κύριος Ντράγκη ότι ανακύπτουν προβλήματα για τις τράπεζες και τη δυνατότητα χρηματοδότησης. Αλλά τελικά θα πρέπει να ε, μιλάμε όχι μόνο για χρηματοδότηση αλλά και για στόχους. Αυτό είναι ζωτική σημασία και το υποστηρίζω. Σε σχέση με τα προγράμματα υπέρ των ε, καταναλωτών, αυτό επίσης ε, προαναφέρθηκε. Θα πρέπει να υπάρχει στοχοθετημένη χρηματοδότηση, γι' αυτό συμφωνώ και επ' αυτού. Επίσης, το, τη σημασία του προγράμματος ε, τελωνίων Μιλάμε για μια κοινή εργασία, τη ραχοκοκαλιά δηλαδή όλου αυτού του σχεδίου ε, πληροφόρησης, επικοινωνίας και τεχνολογιών. Διότι παρά το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν προβλήματα, στο τέλος θα γίνουν πραγματικές οικονομίες που θα είναι πιο αποδοτικές από αυτές που μας είχαν απασχολήσει. Στο παρελθόν είχαμε πολύ δύσκολους τριμερείς διαλόγους. Θα υποβάλω τροπολογίες, αλλά σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι συμβαδίζουμε με την ησυχήτρια και δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Και εγώ θα είμαι σύντομη, φυσικά υποστηρίζω την εισηγήτρια σε ό,τι αφορά το ODR. Προφανώ αυτό είναι πάρα πολύ αναγκαίο, το υποστήριξε άλλωστε και στου κοιόδους εισηγητέ. Υποστηρίζω επίση και το πλωτικό πρόγραμμα. Επί τη ουσία, συμφωνώ με τη γραμμή σα. Το πρόβλημα όμω, όταν εξετάζω πιο συγκεκριμένα τα πράγματα είναι το εξή. Οι επιπτώσει των περικοπών που αποφασίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τι θα σημαίνει στην πράξη. Και θεωρώ ότι στο θέμα των τελωνίων, για παράδειγμα, πραγματικά οι περικοπές θα μας προβληματίζουν. Κοιτάξτε, είναι εμ, αποφάσεις που ελήφθησαν αλλού και εμείς δεν έχουμε παρά να προσπαθήσουμε να τα εφαρμόσουμε τώρα όλα αυτά. Δεν έχουμε κάτι να κάνουμε, αλλά ε, μου προκαλούν κάποια ανησυχία. Γιατί δεν έχει νόημα ουσιαστικά να κάνουμε περικοπές σε αυτούς τους κλάδους. Good. Ωραία. Λέει ο πρόεδρος. Εγώ δεν είμαι επίσημα σκιώδης της ομάδας, αλλά παρακολουθώ το ζήτημα του σύνεγγης και θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτή η χρηματοδότηση μέσα στα πλαίσια και των οικονομιών κλίματος. Θα πρέπει να είμαστε ε, σαφείς με όλη την χρηματοδότηση και να την προωθήσουμε κατά το μέγιστο δυνατό. Ο Λισμίτ είπε ότι θα πρέπει να δεχτούμε το συνολικό πλαίσιο μέσα στα πλαίσια της επανατοποθέτησης. Νομίζω λοιπόν ότι η πλατφόρμα αυτή είναι ύψης της σημασίας. Ως προς τα πιλωτικά σχέδια δεν είμαι και τόσο πεπισμένος. Είδαμε τη, το νέο πακέτο για την οδηγία για τη, τα ταξίδια θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτή η οδηγία ανά το χρόνο. Η κυρία Καρπέλ θέλει να μας μιλήσει για το χρονοδιάγραμμα και μετά θα πρέπει να διακόψουμε. Έχουμε δύο λεπτά μόνο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρο. Πρωτού περάσω στα θέματα χρονοδιάγραμματο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του και συζητητές και για τη συνεργασία αλλά και για τα σχόλια και τι παρατηρήσει του. Σε δύο σημεία θα ήθελα να απαντήσω αν μου επιτρέπετε. Σε πολλά θέματα συμφωνούμε και το σημείο κίνησης ασφαλώ, είναι ότι δεν θέλουμε να γίνουν περικοπές στο δικό μας τομέα αρμοδιότητα. Σε ό,τι αφορά τι διάφορε ε, γραμμέ του προπολογισμού για το 2009 και το 2014 σε ό,τι αφορά και την μελλοντική εξέλιξή τους. Φυσικά η απάντηση και η επεξεργασία των θεμάτων αυτών στην μεμοδότηση θα ήταν κάτι πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο. Έχουμε πλέον μπροστά μας την τελευταία εκδοχή όλων των γραμμών του προπολογισμού και φαίνεται ότι υπάρχει περικοπή 5% σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Αλλά είναι πολύ χρήσιμη η σχετική πρόταση της Επιτροπής. Στους υπόλοιπους συναδέλφους να πω ότι σε ό,τι αφορά τη προσέγγιση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμφωνώ απόλυτα. Έγινε ακρόαση του κ. Τράγκη στην Επιτροπή Οικονομικών Ζητημάτων και σε ό,τι αφορά τη σχετική γραμμή του προϋπολογισμού καταρτίστηκε το σχετικό πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις προτάθηκε 30,8 δισεκατομμύρια και στις πληρωμές μόνο 2 εκατομμύρια. Αυτό τι σημαίνει για μένα ως οικονομολόγος. Φυσικά πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά ως οικονομολόγος τι σημαίνει αυτό για μένα. Ότι έχουμε κάποιο όραμα για το μέλλον, αλλά όχι με συγκεκριμένα στοιχεία, συγκεκριμένο σχέδιο, γιατί δεν έχουμε προβλέψει σχετικές πληρωμές για το μέλλον σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και τα επιπλέον 2,4 δισεκατομμύρια τα οποία θέλουμε να προβλέψουμε, αυτό που προτείνω δηλαδή είναι να προβλέψουμε για τα Ινστιτούτα, για τα Ιδρύματα προτύπων τέτοια αύξηση. Συμφωνώ να διατηρηθούν τα τρέχοντα επίπεδα χρηματοδότησης για τα υπόλοιπα ζητήματα και σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας σε ό,τι αφορά το ODR. Σύμφωνο και με αυτό το θέμα, με αυτά που είπατε. Ξέρω ότι σε ό,τι αφορά το New Europe Travel, σε ό,τι αφορά αυτή την ε, εφαρμογή κινητών δεδομένων, υπάρχουν κάποια ζητήματα. Θεωρώ ότι είναι ωφέλιμη η εφαρμογή αυτή γιατί επωφελεί τον πολίτη και δίνει σε όλο και πιο πολλούς πολίτες την δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσει. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλες τέτοιες εφαρμογές, αλλά αυτή η ευρία εφαρμογή δεν είναι γνωστή δυστυχώς στο ευρύ κοινό. Καλό θα ήταν λοιπόν να είχαμε μια τέτοια εφαρμογή και να μπορούσαμε να τη χρηματοδοτήσουμε με παρκή τρόπο. Ξέρω ασφαλώς ότι έχουμε πολύ περιορισμένα μέσα, αλλά θα μπορούσαμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Το βρήκα και στα έγγραφά μου σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε πολλά τεχνικά ζητήματα να διευκρινίσουμε την Πέμπτη. θα γίνει μια συζήτηση με την ε, αρμόδια Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις σχετικές ε, συζητήσεις και στις 18 Ιουλίου, 12 το μεσημέρι, λίγη προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. 19 Ιουλίου βλέπω στον ε, φάκελο. Ωραία πριν διακόψουμε για το καλοκαίρι. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να το προωθήσουμε γιατί θα πρέπει να ψηφίσουμε μέχρι τις 5 για να μπει στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Ευχαριστούμε την κυρία Γκαλπέλ. Ε, σας ευχαριστούμε όλους και θα τα πούμε στις 3 το απόγευμα για μια ε, διαδικασία για το εμπορικό σήμα, την μεταρρύθμιση, την αναθεώρηση του.